Ε, θέλουμε να ανοίξουμε την πολύ ανοιχτή μας ε, ε, ανοιχτή αγορά και προσπαθούμε να επιτύχουμε τα ευρύτερα συμφέροντά μας στον κόσμο. Όσον αφορά, ε, τα άλλα θέματα, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τα εργαλεία άμυνα, εμπορικής άμυνας και όχι μόνο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα αλλά και απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα μεγάλο κομμάτι της εντολής μας αφορά τη, ε, να, γίνουν, ε, να ανοίξουμε τις αιτήσει για τη θέση του ε, ανώτατου ε, στελέχους που θα ασχολείται με την εφαρμογή των συμφωνιών και Θέλουμε να αντιμετωπιστούν τα εμπορικά εμπόδια, να εξασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας θα, ε, ε, θα ε, τηρούν τις συμφωνίες και θα αναφέρουμε την πρόοδο στην Επιτροπή σας και στα, στους εμπλεκομένους των κρατών μελών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται παράπονα Όλα αυτά θα διατυπωθούν σε ένα έγγραφο πολιτικής που θα δημοσιευθεί και ενδεχομένως μπορεί να συναντηθούμε επ' αυτού. Ελπίζω λοιπόν να ακούσω και τις συστάσεις σας για επ' αυτού. Έτσι, στο πνεύμα αυτό του ανοίγματο και της αμοιβαία συνεννόησης, ε, δεδομένου ότι αυτός είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης, ε, έχουμε προχωρήσει την ε, εμπορική πολιτική χάρη σε αυτά που έκανατε εσείς με την Επίτροπο κυρία Μάλστρομ και θα υπάρχει και δημοσίευση στο διαδίκτυο των αποτελεσμάτων και αυτό που ήταν εποφελές και δημιου... Ε, οικοδόμησε εμπιστοσύνη και προκάλεσε ε, την υποβολή ιδεών. Όλα αυτά θέλω να συνεχιστούν. Γι' αυτό χτες ανακοίνωσα μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες συνεπάγονται ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα ανοίγουν και θα ολοκληρώνουν διαπραγματεύσεις για διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Ε, επίσης, θα προτείνω στο, ε, στην Κομισιόν να δημοσιεύσει περαιτέρω έγγραφα, συστάσεις, ας πούμε, για ε, μελλοντικές διαπραγματεύσεις Επίσης, έχουμε δημοσιεύσει τι συστάσεις για τι διαπραγματεύσει εμπορικών συμφωνιών όπου είναι ε, επικεφαλής οι χώρε. και επίσης έχουμε, θα προτείνω μάλλον, την αναφορά από τις επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις τους. Όλα αυτά στο πλαίσιο της λογοδοσίας και της διαφάνειας και βεβαίως ε, για το, σχετικά με τις μεγάλες ε, επιτροπές ε, εμπορίου της άμυνας, εμπορίου άμυνας. Υπάρχουν φυσικά ε, και διαπραγματεύσεις που υπάρχει εμπιστευτικότητα, αλλά γενικά πιστεύουμε ότι η κοινή γνώμη πρέπει να, είναι, να γνωρίζει πώς εφαρμόζονται οι δίκες πρακτικές και ο ανταγωνισμός. Θα στηρίξω και τις πρωτοβουλίες για τον κανονισμό για τη διαφάνεια. Αυτές είναι κάποιες από τις ιδέες που ανακοίνωσα ήδη, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί η διαφάνεια. Πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση με τον κόσμο. Η πρόσφατη παράμετρος δείχνει ότι υπάρχει υποστήριξη για το εμπόριο, αλλά υπάρχουν και αμφιβολίες ε, και φόβοι. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό, είναι ευθύνη μας. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να, υπάρχουν, να έχουμε διαλόγους σε άλλες εκδηλώσεις. Έχω δει κάποιο ενδιαφέρον υλικό του Κοινοβουλίου σχετικά από μαρτυρίες, ταινίες κλπ. Και από τους Ευρωβουλευτές και από το θεσμικό όργανο. Πρόεδρε, Αυτά ήθελα να παρουσιάσω και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Perfect, Commissioner. τον Επίτροπο. Additional good news. Για τη διαφάνεια είχαμε και άλλα καλά νέα. Είμαι πεπισμένος και είμαστε πεπισμένοι ότι η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει στήριξη για την εμπορική πολιτική. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες καταρχήν για τέσσερα λεπτά έκαστος. Ο, το έλκυνε πρώτος, ο κύριος Μπόμαν. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Warborn. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε στην Επιτροπή μας σήμερα. Το ερώτημά μου αφορά τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ΠΟΕ. Καταρχά, μπορείτε να μα ενημερώσετε για τι διαπραγματεύσει και το γύρο διαπραγματεύσεων που έλαβε χώρα συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι πρόοδο σημειώθηκε, τι κάνει η Κομισιόν αυτή τη στιγμή και πώς θα χρησιμοποιήσετε το χρόνο σας ε, μέχρι την Υπουργική Σύνοδο. Μπορείτε να μας πείτε επίσης δύο λόγια για τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας και αν μπορούν να μας πούν κάτι για το πώς θα προχωρήσουμε στον επόμενο διαπραγματευτικό γύρο. Είναι προάγγελος ε, κάποιων αλλαγών. Μια και είναι πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις ε, ροές δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Πάντα για το ίδιο θέμα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και πώς συνεργάζεται με τους άλλους επιτρόπους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κάτλιν Φαν Μπρέντ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητές σας και της Επιτροπής ΙΝΤΑ, της Επιτροπής μας. Θέλω να μιλήσω για την εφαρμογή, για την πιθανή σύμφωνη γνώμη και πιθανές νέες εμπορικές ε, συμφωνίες. Όλα αυτά μαζί. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα στην Ολλανδία κάνουμε συζητήσεις για την έγκριση της ΣΕΤΑ. Γράψατε μια μακροσκελή επιστολή στην Ολλανδική κυβέρνηση και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και δύο πράγματα μου τράβηξαν την προσοχή και είναι σημαντικά για το μέλλον, νομίζω. Και τα δύο αφορούν την ουσία της συζήτησης. Καταρχάς, οτιδήποτε συνδέεται με θέματα προστασίας ε, των επενδύσεων από το ISDS έως το ICS. Και στην Ολλανδία και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν πολλές ανησυχίες γιατί, για το πώς λειτουργεί το επενδυτικό αυτό δικαστήριο. Είπατε ότι θα είναι διαφανές δικαστήριο με αρμόδιους ε, ε, δικαστές, ε, διαφάνεια, ε, διαφανείς διαδικασίες και προσπελάσιμο στην κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον. Το δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά τους δικούς μας κανόνες. Για το βόλιο, Φερρυπίν. Ε, για το βόλιο με ορμόνες. Τους κανόνες μας. Θέματα που τα διαβάσαμε σε πολλά σε πολλέ εφημερίε αυτή τη βδομάδα για τα φυτοφάρμακα, τα οποία είναι απαγορευμένα ή εν μέρει απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπαίνουν μέσω των εμπορικών σχέσεων προϊόντα με φυτοφάρμακα και φτάνουν στην αγορά μα και μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν φτάνουν στο ύψο των δικών μα προτύπων. Το ίδιο και για το κλίμα. Είπατε κάτι σημαντικό στην επιστολή σα. Ξέρετε ότι είναι σημαντικό κατά την άποψή μα αυτά τα κεφάλαια να εφαρμόζονται και να υπάρχουν και κυρώσεις. Να υπάρχουν κυρώσεις σε αυτά τα κεφάλαια. Πρέπει να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αλλιώς θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο όλες οι μελλοντικέ ε, συμφωνίες ελευθερού εμπορίου να τις προσυπογράψουμε. Είπατε για τη TST και την εφαρμογή της. Είπατε ότι μπορεί να γίνουν ε, αλλαγές στην πολιτική και κατά πόσο το θέλουμε αυτό. Πρέπει να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς το κεφάλαιο αυτό θα γίνει πιο εκτελεστό και θα βασίζεται και θα υπάρχουν και κυρώσεις εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Η Karen Κράτσπορ από το Renew. Μόλις πέρασε η συμφωνία για το Βιετνάμ με πλατιά πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ήταν σαφής δήλωση υπέρ του ελεύθερου και βιώσιμου εμπορίου αυτή η στάση μας. Χαίρομαι γι' αυτό. Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε καλές δεσμεύσεις εν ώψη της ψηφοφορίας και η πλατιά πλειοψηφία δείχνει ότι είμαστε σε θέση να παίξουμε παγκόσμιο ρόλο στο εμπόριο Μας περιμένουν πολλά σημαντικά πράγματα μπροστά μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παρακολούθηση αυτής της συμφωνίας, πρέπει να την παρακολουθήσουμε το ή άλλως. Ποιος είναι ο ρόλος το, του νέου επικεφαλής ε, για θέματα εφαρμογής. Ποιο είναι ο ρόλο του κατά απόψη σα, πώ τον βλέπετε. Για την Κίνα, επίση, δεύτερο θέμα. Ο, πρέσβης ο πρέσβη τη Κίνα στη Σουηδία απείλησε ότι η Κίνα θα επιβάλλει ε, εμπορικούς περιορισμούς στη Σουηδία. Όταν ο Υπουργός ε, ε, Πολιτισμού έδωσε στην ήμαν η οποία είχε κρατηθεί χωρίς δίκη από τις Κινέζικες Αρχές για τέσσερα χρόνια, βραβείο. Είναι πολύ περίεργο νομικά αυτό να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τι σκέφτεστε ότι μπορεί να γίνει. Πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο. Γιατί αυτές οι απειλές είναι απαράδεκτες. Τρίτη ερώτηση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Το μηχανισμό προσαρμογής των σύνορων στο θέμα του άνθρακα, του διοξείδιο του άνθρακα δηλαδή. Ε, μιλάμε για, τον αγώνα κα, κατά της κλιματικής αλλαγής. Είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε αυτό το θέμα με άλλες χώρες, με άλλες περιφέρειες. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες παγκόσμια, άλλες χώρες οι οποίες έχουν ε, παρόμοιες ιδέες. Ο Καναδάς, Φερρυπίν θα μπορούσαμε να βρούμε εταίρους και να συνεργαστούμε μαζί τους ε, για να καταπολεμήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο την ε, αλλαγή του κλίματος. Ευχαριστούμε για την ID ο κύριος Ζουδά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε και θα αποτιμούσα να μιλήσω γαλλικά, αν δεν σας πειράζει. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι συνολική και πολύ προσωπική για τον Επίτροπο. Δεν φοβάστε μήπως σύντομα βρεθείτε εντελώ μόνος. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με εκπροσώπους του Φόρουμ για τις χώρες της Ασίας και μου είπαν κάποιους αριθμούς. Σήμερα το 2, τα δύο τρίτα του ΑΕΠ παγκοσμίω και του παγκόσμιου πληθυσμού ανήκουν σε κράτη που, προσ επιδιώκουν να προσπιστούν τα εθνικά του συμφέροντα με τρόπο μάλιστα ε, αυστηρό και έντονο και κοιτάζουν ε, τα δικά του εθνικά συμφέροντα να περάσουν πάνω απ' όλα. Ε, δεν λέω ότι είναι εθνικιστέ, αλλά είναι πολύ ρεαλιστέ σε εθνικό επίπεδο. Και λίγοι ενδιαφέρονται για την πολυμερή προσέγγιση και γενικώ για τα θεσμικά όργανα τη πολυμερού προσέγγιση. Η ερώτησή μου λοιπόν, ενώ παντού στην Ευρώπη ο κόσμο αρχίζει να είναι όλο ένα και λιγότερο ευνοϊκό σε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών ε, στην Ευρώπη και νομίζω ότι η επιδημία από την Κίνα το δείχνει αυτό εύκολα. Ε, η, πέρα από την απελευθέρωση του εμπορίου, έχουμε τώρα και κινδύνου για το περιβάλλον και την υγεία. Ο κόσμο αρχίζει να πιστεύει ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μετατοπίσουμε στη δική μα την ήπειρο τι δραστηριότητέ μα και στα δικά μα τα κράτη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλούστατη δεν αισθάνεστε λίγο απομονωμένο, λίγο μόνο. Ποιοι θα είναι οι συμμαχοί σα για να αναθεωρήσετε και να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του ΠΟΕ, ε, να ε, ξεκινήσει σε, ένα καινούριο, σε μια καινούργια βάση και να προχωρήσουμε σε πολυμερεί συμφωνίε. Και επίση μια ερώτηση κάπω ε, πρακτική, λειτουργική. Τη λέω Γάλλο. Άκουσα προηγουμένω ότι οι διευθυντέ μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία θα είναι στην έκθεση των γεωργικών προϊόντων για να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους προς τους ε, γεωργούς της Γαλλίας και τους κτηνοτρόφους ε, σε σχέση με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΙΠΑ, τις οποίες τις έχουν υπολογίσει πάρα πολύ καλά οι Αμερικανοί για να διχάσουν τους Ευρωπαίους, να τους βάλουν τους μεν ε, να βρίσκονται στην παλότητα με τους δε και στον οικονομικό τομέα, στη γεωργία αλλά και στην αεροναυπηγική θέλουν να μας τρέψουν τους μεν εναντίον των δε. Εδώ λοιπόν πολύ πρακτικά ποια στρατηγική, ποια λύση μπορούμε να προκρίνουμε για να ξεπεράσουμε τους διχασμούς μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και να μην έχουν αντιπαλότητα μεταξύ τους οι διάφοροι μηχανικοί κλάδοι της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ και για τους πρασίνους η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Νομίζω αυτά που μας είπατε ήταν ευχάριστες ειδήσει για τη διαφάνεια. Να συνεχίσετε και να ενισχύσετε την πολιτική του προκατόχου σας που είχε διευρύνει τι διαπραγματευτικές εντολές για να τις γνωρίζει και το κοινό και να ξέρουν τι συζητάμε. Εγώ όμω κάπω έχω εκπλαγεί με ένα από τα εμβληματικά, με τι εμβληματικέ αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πράσινη Συμφωνία. Διότι είναι σημαντική η εξωτερική τη ε, διάσταση και είναι πολύ μετριοπαθή η πρωτοβουλία ω προ την εμπορική πολιτική. Οι υπηρεσίε σα λοιπόν έχουν συνεννοηθεί, έχουν συντονιστεί ώστε η εμπορική μα πολιτική να συνάδει με τι επιταγέ τη Συμφωνία των Παρισίων και να είμαστε και βέβαιοι ότι στο μέλλον θα έχουμε και καρπού στι διαπραγματεύσει μα ε, με τι άλλε χώρε και τι άλλε γεωγραφικέ περιοχέ, Εκεί όπου ε, η Συμφωνία των Παρισίων είναι δεσμευτική και για του μεν και για του δε. Επίση, να ρωτήσω για την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική. Ε, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε πότε αυτή η ανακοίνωση θα συμπεριλαμβάνει πτυχέ που έχουν να κάνουν με τη διεθνή εμπορική πολιτική τη Ένωση το βλέπετε ως μια ευκαιρία, αν συμβεί αυτό, να διασυνδέσουμε τη μηχανική πολιτική με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην εξωτερική διάσταση τουλάχιστον. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για την δέους επιμέλεια, για τις αλλαγές, την ενεργειακή ένταση ε, και άλλα παρόμοια ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για του εσωτερικού μεταρρυθμιστέ, ο κ. Μπουζουά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για την ε, παρουσίασή σα και νομίζω ε, συμμεριζόμαστε τι φιλοδοξίε σα. Θέλουμε ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ιδίω σε αυτού του καιρού, ε, του ταραχώδει, του καιρού βεβαιότητα και στάθεια. Συμφωνώ χρειαζόμαστε το εμπόριο και θα πρέπει να διέπεται από κανόνες. Βεβαίως, η πολυμερής προσέγγιση είναι σημαντική, να διασώσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, βεβαίως, αλλά για τα μονομερή μέτρα των ήπα βλέπω ότι κάποιες φορές έχουν και κάποια βάση ως προς το κόστος της διαδικασίας, ως προς αυτό που ονομάζουν την ε, ανεξέλεγκτη εξουσία των δικαστών ε, εδώ πρέπει να δούμε τι κανόνες εγκρίνονται ε, σε τοπικό επίπεδο ε, και σε καιρούς ηλεκτρονικού εμπορίου, σε καιρούς κανόνων για το περιβάλλον. Τι προοπτικές βλέπετε εσείς για να φτάσουμε σε μια συμφωνία και να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον, το πολυμερές, τους οργανισμούς με πολυμερή προσέγγιση και να βρούμε διέξοδο στη, στα σημεία που έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Επίσης, θα πρέπει να αναζητήσουμε συμφωνία σε κάποια σημεία με, την, με τη ΣΥΠΑ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι σαφές αυτό, γεωπολιτικά αυτό πρέπει να επιδιώξουμε και είναι σημαντικό για πολλέ από τι προτεραιότητε μα. Τι προοπτικέ όμω διαβλέπετε εσεί συγκεκριμένα ω προ την Κίνα. Δεν πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι κανόνε παιχνιδιού, ε, ίσοι όροι και θα πρέπει να δοθεί τέρμα στην μεταφορά τεχνολογίας και τις κρατικές επιδοτήσεις. Να υπάρχει ίσως ανταγωνισμός για την Ινδία. Σημειώνω ε, την επιφυλακτικότητά σας. Ε, πιστεύετε όμως ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε κάποιο είδους συμφωνία, έστω και εν μέρη συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο. Ισω μια συμφωνία προστασία των επενδύσεων τουλάχιστον. Διότι έχουμε 22 διμερεί συμφωνίε με 22 κράτη-μέλη της Ένωσης. Ε, δεν υπάρχει προστασία για τις επενδύσεις και δεν είναι δυνατόν να... Μήπω είναι δυνατόν να φτάσουμε σε συμφωνία προστασία των επενδύσεων. Πραγματικά είμαι υπέρμαχο αυτή τη επιλογή. Και ε, τέλο, για τις εντάσεις που είδαμε να προκύπτουν από την διαδικασία έγκριση των συμφωνιών μας με το Βιετνάμ και τον Καναδά. Βλέπουμε ότι για το σύστημα διευθέτησης ε, διαφορών με επενδυτές σε δικαστικό επίπεδο ε, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχει κώδικα συμπεριφοράς, ανεξάρτητοι δικαστέ, καλύτερη πρόσβαση για τι σε κάποιε χώρε είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθεί κανεί σε τοπικά δικαστήρια. Οπότε, μακροπρόθεσμα, ίσω ένα τέτοιο σύστημα να ήταν η καλύτερη λύση. Πολυμερέ δικαστικό σύστημα. Ευχαριστούμε και για την ΚΟΕ ο κύριο Σόλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, Επίτροπε, για τα πολύ ξεκάθαρα λόγια σα σε ό,τι αφορά τη διάσταση τη διαφάνεια. Διαβεβαιώ ότι από την πλευρά τη δική μου ομάδα θα έχετε όλη τη στήριξη που χρειάζεστε για τι διαβουλεύσει και τι συζητήσει με του πολίτε για την εμπορική πολιτική να γνωρίζουν γιατί διαπραγματευόμαστε και σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδεύσουμε στον 21ο αιώνα. Και ε, έρχομαι έτσι στην πρώτη μου ερώτηση. για τις είπα, τα μέσα μαζικής ενημέρωση λένε ότι προτείνεται συμβαστική συμφωνία στις ΕΠΑ που καταργούν μερικούς βασμούς ε, σε γεωργικά προϊόντα με μηδενική βασμολογική ε, επιβάρυνση στα αλλιευτικά και και σε κάποια ακόμα βιομηχανικά προϊόντα. Μπορείτε να μας πείτε αν ισχύει και θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτή η συμφωνία από την εντολή σας. Πώς να τις αντιληφθούμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, πού το πάτε. Ε, διότι είναι κρίσιμα τα πράγματα για το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και πολλά άλλα στις εμπορικές σχέσεις όπως με τις είπα. Για την Κίνα το έθιξαν και άλλοι συνάδελφοι. Είναι μεγάλη πρόκληση, είναι μεγάλη δυσκολία για μας δεν λέω βεβαίω ότι το ICT, το σύστημα το δικαστικό για του επενδυτέ, είναι το μόνο που θα καθορίσει τι εμπορικέ μα σχέσει. Ο κόσμο καταναλώνει. Οι εμπορικέ σχέσει συνάπτονται αυθορμήτω. Ε, και πρέπει να υπάρχουν κριτήρια βιωσιμότητα. Εδώ λοιπόν η ερώτησή μου είναι, αναμένεται πολιτική συμφωνία στην ε, ε, συζήτηση για την πρόσβαση των επενδυτών στην αγορά. Και αυτή η συμφωνία θα συμπεριλαμβάνει δεσμεύσει που θα φτάνουν στο επίπεδο του, Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία ανάλογα με αυτά που περιέχει η συμφωνία με το Βιετνάμ. Και όπω ήδη αναφέρθηκε. Η ερώτηση είναι πόσο ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της ε, βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι η στόχη της χιλιετίας ε, ένα ορόσημο. Η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ένα ορόσημο δίκτυς συγκριτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε για να προχωρήσουμε. Ε, και έχουμε και το σύστημα της κυκλικής οικονομίας με το κεφάλαιο TFT πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι αντικείμενο εμπορία ε, και πώ θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μα με τρίτε χώρε. Πρέπει να δούμε ε, εάν θα υπάρχει δυνατότητα παραγωγή και πώ το εμπόριο θα μπορεί να ε, έχει και κάποιο μέλλον. Ευχαριστώ. Εγώ από πλευρά μου θέλω να κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε τον πρώτο γύρο. Το σημείο 3 της δουλειάς που σας βάλαμε για το σπίτι είναι το το θέμα της δέουσας επιμέλειας και της εμπλοκής της είναι εφοδιαστική αλυσίδα. Ε, ε, από πλευράς Κοινοβουλίου και Συμβουλίου υπάρχει το θέμα της νομοθετικής στήριξης για, την, ε, για νομοθέτημα δέουσας επιμέλειας. Έχετε ιδέες για το πώς θα γίνει αυτή η εμπλοκή σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κύριος Βόρμπαν ρώτησε για την πρόοδο που σημειώνεται. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσιεύτηκε μια νέα στρατηγική δεδομένων που θα μας ενημερώσει και για την ε, ε, διαπραγματική μας θέση για το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ΠΟΕ. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, θέλει να είναι κυρίαρχη η Ένωση επ' αυτού, αλλά αναγνωρίζουμε ότι οι ροές δεδομένων πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, αλλά και δεν υπάρχουν σύνορα. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία στην Ένωση, λόγω του τεράστιου όγκου ε, βιομηχανικών δεδομένων, τα οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα και άρα είναι ευκαιρίες θέσεων εργασίας. Στον ΠΟΕ αυτό το οποίο κάνουμε συγκεκριμένα είναι να υποβάλουμε προτάσεις στις διαπραγματεύσεις που διευκολύνουν τις ε, επιγραμμικές ε, συναλλαγές, διαδικτυακές συναλλαγές, τις υπογραφές Επίση, κανόνε που στοχεύουν στην ενίσχυση τη εμπιστοσύνη των καταναλωτών διαδικτυακά, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, ε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι και να πει κανεί ε, σε σχέση με αυτά που λέει ο κύριο Facebook. Το Facebook τουλάχιστον αναγνώρισε τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ε, ιδιωτικότητα. Προσπαθούμε να υπάρξει να ασχοληθούμε την ε, μόνιμη απαγόρευση των ηλεκτρονικών μεταβιβάσεων διαφόρων βίντεο κλπ. Αυτά είναι απλά παραδείγματα ε, σε σχέση με τους στόχους μας και συγκριτικά με άλλους. Προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις αυτές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και εμείς συνεργαζόμαστε στενά. Είναι ένας από τους λίγους τομείς που είμαστε σε στενή συνεργασία, αλλά εδώ ε, συμφωνούμε, θέλουμε να υπάρχει ισότητα ευκαιριών, εμπιστοσύνη του καταναλωτή και να εξασφαλιστεί ότι η ίδια η Ένωση δεν θα πληγεί από θέμα που θα αφορά την, τον, το, το, ε, τοπικότητα, την, τον εντοπισμό των δεδομένων. Υπάρχουν θέματα ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό θέμα. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα ολοκληρώσουμε τα θέματα ε, μέχρι το τέλος Ιουνίου στον Ουσουλτάν, αλλά ελπίζουμε ότι θα υπάρχει κάποιο κείμενο. Και αν επιτευχθεί αυτό, θα σημάνει ουσιαστική πρόοδο. Ενδεχομένως μπορεί να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο τέλος του χρόνου. Αυτό ελπίζει η Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι εδώ. Τα, το έγγραφα που δημοσιεύθηκαν σήμερα θα ενημερώσουν την πράξη των ε, ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως ακούσατε και από κάποιον άλλον, υπάρχει αυτό και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουμε, ανάλογα με το ρυθμό που θα επιτευχθεί βέβαια. Κάτλιν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ε, ήμουν σε επαφή με τις αρχές ε, στην Ολλανδία και προσπάθησα να διευκρινίσω κάποια θέματα παραπληροφόρησης που υπήρχε. Δεν προτείναμε καμιά αλλαγή, απλώς ξεκαθαρίσαμε τα συμφωνηθέντα. Μερικές φορές οι άνθρωποι μελετούν τις συμφωνίες και άλλες δεν, το, δεν τις μελετούν και τότε ζητούν από την Επιτροπή να δώσει διευκρινήσεις και το κάνουμε. Δεν θέλω να ε, προλάβω τι θα πει αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα λέω ότι ε, έχουμε προσδοκίες. Είναι δύσκολο να υπάρξει θετική ψήφος στη ΣΕΤΑ, αλλά τελικά εγκρίθηκε ε, με τρεις ψήφους, πολύ μικρό ε, μικρό περιθώριο. Όλες οι νίκες στην Ολλανδία γίνονται με μια μικρή διαφορά. Πάντοτε η χώρα αυτή όμως μας υποστήριζε τους ανοιχτούς κανόνες των διεθνές εμπόριων είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον τομέα των εξαγωγών. Δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας, εργασίας στις Ολλανδίες. 160 δις, ε, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πριν πέντε χρόνια. Η Ολλανδία είναι ένας από τους ηγέτες στο εμπόριο και στην βιωσιμότητα του εμπορίου. Και αυτό έχει αναγνωριστεί. Το καναδικό σύστημα σε σχέση με το ICS είναι πολύ ενδιαφέρον δείχνει τι θέλουμε να πετύχουμε σε σχέση με τη συμφωνία με τον Καναδά και φυσικά αυτό το δοκιμάζουμε, να δούμε αν θα λειτουργήσει. Θα συναντηθώ με τις αρχές του Καναδά στις επόμενες δύο εβδομάδες για να το συζητήσουμε στις περισσότερες λεπτομέρειες στο σύστημα. Υπάρχει και το θέμα της κοινωνίας των πολιτών που πρέπει να ενημερωθεί με διαρθρωμένο τρόπο. Συμμερίζομαι την αρχική, τη θέση αρχής που έχετε. Το θέμα των ε, φυτοφαρμάκων που αναφερθήκα, το οποίο αναφερθήκατε σε τρίτες χώρες, το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, το θέμα των φυτοφαρμάκων. Αλλά ή η προσέγγιση μας στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία είτε όχι. Υπάρχει διάσταση απόψεων από αυτόν. Εγώ ε, είμαι υπέρ της χρήσης της επιστήμης. Οι αγρότες θα πρέπει να έχουν τις σωστές εναλλακτικές γιατί μιλάμε για την υγεία των πολιτών. Είτε η απαγόρευση είτε όχι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια ο, κύριος, ο Επίτροπος Κυριακίδης και η όλη η αγροτική στρατηγική θα πέσει σημαντικό ρόλο στη διατύπωση της άποψης Κομισιόν για το θέμα αυτό στο άμεσο μέλλον. Νομίζω μέχρι τέλος Μαρτίου θα δούμε προτάσεις. Η ασφάλεια του καταναλωτή ήταν και πάντοτε θα είναι μια σημαντική ε, αρχή για μας. Με βάση βεβαίως ε, τα ευρήματα της επιστήμης. Κάνουμε διαπραγματεύσεις και έχουμε προχωρήσει στην παραγωγή αυγών. Στη συμφωνία με τον, τις χώρες Μερκοσούρ ζητήσαμε διευκρίνηση και επαλήθευση σε σχέση με την παραγωγή των προϊόντων. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουμε και σε άλλα προϊόντα έτσι στο μέλλον. Δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω τι θα πει ε, η συνάδελφος Κυριακίδη. Το, η τροφή των Ευρωπαίων είτε θα είναι χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή θα έχει τα νόμιμα υπολείμματα. Νομίζω όλοι θέλουν να είναι όσο πιο φιλόδοξοι γίνεται. Τι και οι κυρώσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία εδώ, ε, στο σώμα αυτό, ε, σε σχέση με τις κυρώσεις. Αν βάλετε τις κυρώσεις επιτάπητος, θα υπάρξει δυσκολία στη συμφωνία. Εντάξει, αν αυτό επιθυμείτε αλλά είναι μια ανοιχτή άποψη, είμαι στα χέρια σας σε σχέση με αυτό που θέλετε να κάνετε. Η εμπειρία μου μου έχει διδάξει όμως ότι όταν επιδιώκεις ε, την αρχή της ε, προφύλαξης, τη συμφωνία του Παρισιού, κυρώσεις, το τίμημα το πληρώνουμε κάπου αλλού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Βεβαίως συμφωνώ να πετύχουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε σε σχέση με το TST. Τώρα, ε, ο ρόλος ε, του Chief Trade Enforcement Officer. Υπάρχουν κάποιες αρχές ε, τις οποίες θα δημοσιεύσουμε και θα το συζητήσετε για να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος, να είναι ουσιαστικός και να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε όντως θα συμβεί. Οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι, παραδείγματος χάρη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίρνουν μόνο το 35% της αξίας του ωφέλους του ε, εμπορίου των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Πρέπει αυτό να βελτιωθεί. Πρέπει να υπάρχουν ε, ε, εργαλεία να βελτιώνουν το όφελος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι το 80% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν περισσότερο από τις ε, συμφωνίες ελευθεροπορίου και να, η βοήθεια θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Να δοθούν περισσότερα στις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Άρα πρέπει να ανακοινώσουμε πιο ξεκάθαρα τι θα απαιτηθεί από αυτή τη θέση. Δεν ήξερα ότι η Σουηδία απειλείται από τους Κινέζους. Ίσως θα μπορέσετε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες και με τα χαράς θα ε, παρακολουθήσω το θέμα αν με ενημερώσετε. Όσον αφορά τον μηχανισμό, ε, μεθοριακό μηχανισμό άνθρακα, Θέλω να αποφύγω να χρησιμοποιήσω τη λέξη φόρος, σε μπάση περιπτώσει. Πρέπει, όπως είπαμε, να είναι συμβατός με τον ΠΟΕ. Όρο και αυτό εδώ είναι ένα θέμα. Υπάρχουν διάφοροι κανόνες για το πώς πρέπει να είναι ε, αυτός ο μηχανισμός. Ο Επίτροπος Μπιζεντιλόνη προχωρεί αργά για να, κάνει, να προχωρήσει καλά. Δεν περιμένω ε, πρόταση πριν από τα μέσα του επόμενου έτους. Δεν θέλουμε να βλάψουμε κατά λάθο τη βιομηχανία μας, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε επίση ότι θα υπάρχει μια τιμή του άνθρακα και ότι το ευρωπαϊκό Green Deal ε, βοηθάται σημαντικά από αυτή, αυτό το μηχανισμό. Δεν ξέρουμε αν θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς ή άλλους κλάδους. Ο κύριος Τζεντιλόντι θα το συζητήσει με ανοιχτό μυαλό. Και αυτός είναι πολύ καλή, καλός τρόπος να ξεκινήσει κανείς. Ενδεχομένως μπορείτε να τον καλέσετε να συζητήσετε. Δεν αισθάνομαι μοναξιά ως Επίτροπος Εμπορίου. Έχουμε 31 εμπορικέ συμφωνίες σε, 17, σε 70 χώρες. Ε, είναι καλό αυτό. Ουσία παρά ταχύτητα. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία επενδύσεων με την Κίνα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα, τι θα πετύχουμε. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, βιομηχανικών επιδοτήσεων έτσι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι σε μειονεκτική θέση ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και και υπάρχει τώρα και μια νέα φράση, η ισότιμη, ισότιμη βάση στο εμπόριο. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπάρξει ισοτιμία, είτε μιλάμε για τις επιδοτήσεις, είτε το περιβάλλον, δικαιώματα εργαζομένων, τα θέματα πρότυπα τροφίμων κλπ. Έχω αρκετούς υποστηριχτές στον ΠΟΕ, με τα χαρά στο ακούω, σε σχέση με όλα αυτά υπάρχουν 16 κράτη-μέλη που έχουν προσυπογράψει την μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και το πολυμερές σύστημα που προσπαθούμε να ε, θεσπίσουμε σε σχέση με την κατάρρευση του ε, συστήματος υποβολής προσφυγών, του οργάνου των προσφυγών. Θα γίνει μια συνάντηση της ε, ομάδας ΟΤΑΒΑΣ στις 18 Μαρτίου θα γίνουν και οι συναντήσεις του ΟΣΑ με τα θέματα αυτά το Μάιο για να δούμε αν θα προχωρήσουμε πριν από τη συνάντηση του Νου Σουλτάν τον Ιούνιο. Έτσι προσπαθούμε να έχουμε ηγετική θέση όσο πιο καλά μπορούμε. Για τους αμερικανικούς ε, δασμούς και την Airbus, η Airbus είναι γαλλική εταιρεία, αλλά έχει δορυφορικές εταιρείε σε διάφορα άλλα κρατημέλη και υπάρχουν 22 άλλα κρατημέλη τα οποία επηρεάζονται από τους δασμούς λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτό το πάνελ για την Airbus του ΠΟΕ. Βοηθάμε λοιπόν την Airbus, δεν, είναι το αντίθετο, δεν γίνεται το αντίθετο. Συνεργαζόμαστε και λόγω του, της ε, περίπτωσης του Airbus έχουμε αυτή τη διαμάχη με τους Αμερικανούς. Ε, πριν από καμιά δύο εβδομάδες στην Αμερική προσπάθησα να κάνω μια διπραγματευτική διευθέτηση για την Airbus. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε στον ΠΟΕ, αλλά οι φίλοι μας οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δεν θα έχουμε το ίδιο επίπεδο κυρώσεων ε, για την Boeing όπως με την Airbus. Ίσως κάνει λάθος. Και κατά πολύ λάθος. Αλλά από εδώ μέχρι τον Ιούνιο ε, προτιμώ να διαπραγματευτούμε και για την Airbus και για την Boeing και θέλω ε, και οι δύο εταιρείες να συμμορφωθούν και να εξαλειφθούν οι δασμοί. Την περασμένη Παρασκευή ε, υπήρχαν πολλές προσδοκίες στον τύπο έξαρση, έτσι, ότι θα υπήρχε τρομερή αύξηση των δασμών και ότι θα προσταθούν και άλλα προϊόντα, αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι καλό. Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα που έστειλαν οι Αμερικανοί. Ότι θέλουν δηλαδή να συνομιλήσουν μαζί μας σοβαρά για να συνοηθούμε για αυτά τα θέματα. Ελπίζω να μην είμαι αφελής. Ε, ειλικρινά, θεωρώ ότι έχουμε ευκαιρία την καλύτερη ευκαιρία που είχαμε το τελευταίο διάστημα να, να, αντιμετωπίσουμε το θέμα των δασμών ε, για το Airbus και το κρασί των Γάλλων. Επίσης, ε, το 1ο Νοεμβρίου μπήκαν οι δασμοί, μέχρι τότε είχαμε πολλές εξαγωγές. Ε, από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ας πούμε, οι εξαγωγές της Γαλλίας προς την Αμερική μειώθηκαν. Ε, γιατί όμως και γιατί το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ε, εξήχθηκαν πάρα πολλά προϊόντα. Το συνολικό νούμερο είναι 1% αύξηση. Θα μιλήσετε σε λίγο, περιμένετε. Έχω τα νούμερα. Συνολικά τα νούμερα τι λένε. 1% αύξηση για το 2019 συνολικά. Έτσι. 1% αύξηση. Πήγαν απάνω, ανέβηκαν οι εισαγωγέ. Οι Γάλλοι μα λέγανε ότι θα ήταν λιγότερε. Δεν έγινε αυτό. Ε, αντίθετα, ανέβηκαν οι εισαγωγές. Για το, τη Συμφωνία του Παρισιού και την Πράσινη Συμφωνία είπαμε ότι οι συνολικές εμπορικές ε, συμφωνίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τη Συμφωνία του Παρισιού. Θα είναι ουσιαστικό κομμάτι αυτών των συμφωνιών. Στην, εμπορικά, στην εμπορική, πολιτική θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάθε πτυχή της ζωής ε, και το ίδιο γίνεται και στην Πράσινη Συμφωνία στην ε, βιομηχανική στρατηγική προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και στην ψηφιακή στρατηγική. Όλα, όλες αυτές οι συμφωνίες στηρούμε τις αρχές από τις οποίες διέπεται η Πράσινη Συμφωνία. Κύριε Μπουζουά, νομίζω ότι αρκετά μίλησα για τον ΠΟΕ. Είμαστε, κάνουμε μια προσπάθεια στην πολυμέρεια, ε, η οποία βασίζεται στους κανόνες. Είναι το DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα και τι ΗΠΑ να τι δω να συζητάνε μαζί μα αυτά τα θέματα που μα ανησυχούν. Αλλά πρόσφατα είχαμε αυτό το πρόβλημα με το σώμα προσφυγών, το μελετήσαμε την περασμένη ε, Τρίτη. Κάποιε από τι ιδέε ε, που αναφέρουν οι Αμερικανοί, τι συμμερίζομαι, ότι θέλουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική οργάνωση. ΠΟΕ δηλαδή. Έχουμε 164 χώρε. Ε, αν θέλουμε να συνοηθούμε 164 χώρε και να φτάσουμε στη συνένεση, ε, πολύ δύσκολο είναι αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει η πολυμέρεια, ότι είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες. Ε, επίσης, ε, συναντήθηκα με την Ινδία για θέματα ε, εξωτερικών υποθέσεων. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει συμφωνία ελευθερών με την Ινδία στο εγγύς μέλλον. Ε, το 2013 αναστήλαμε τις σχέσεις μας και δεν νομίζω ότι έχουν οριμάσει συνθήκες για να αλλάξουν τα δεδομένα. Αν όμως ε, μας κάνουν κάποιες προτάσεις, και μας δώσουν λόγο να αλλάξουμε τη στάση μας και να κάνουμε πρόταση, γιατί όχι, θα εξετάσουμε. Αλλά όπως είπα και στην Κάτλιν Βαν Μπρέμ, το σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα, ούτω ώστε να ε, διορθώσει τα κακό κείμενα. Κύριε Σούλτς, οι προτάσεις ε, των Αμερικανών δεν εκφεύγουν τη σημερινή εντολή. Δεν θα πρέπει να πιστεύετε ότι λένε οι εφημερίδε σε σχέση με αυτά που προσπάθουμε να κάνουμε. Όταν σας λέω ότι είναι εντός της εντολής, σημαίνει ότι έχουμε και ένα πιο, μια πιο στενή περίμετρο για να κινηθούμε απέναντι στους Αμερικανούς. Ε, στα υγειονομικά και φυτογειονομικά θέματα έχουμε προχωρήσει κάτι, κάπως, αλλά δεν συμφωνούμε. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε καμία περίπτωση να μειώσουμε και να κατεβάσουμε τα πρότυπά μας. Ε, για το περιβάλλον, ε, τα πρότυπα για τα τρόφιμα. Έχουμε μια περιορισμένη εντολή και εντός αυτής δουλεύουμε. Και εντός αυτής θα συνεργαζόμαστε και θα συνομιλούμε με τους Αμερικανούς. Τώρα, για το αν θα φτάσουμε συμφωνία με τους Κινέζους το Σεπτέμβριο, δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη αυτή τη φάση, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα λόγω κοροναϊού. Πολλές συνεδριάσεις ακυρώθηκαν ε, θα πρέπει λοιπόν λόγω της συνόδου της ε, λειψίας να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τον ε, Ιούλιο. Εσύ προχωρούμε για πολλά θέματα με τους Κινέζους, για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και μεταφορά τεχνολογίας. Εκεί έχουμε κολλήσει λιγάκι, δεν συμφωνούμε. Δεν θέλω να σας πω ότι έχουμε, δεν κάνουμε καμία πρόεδρο. Για πολλά θέματα έχουμε προχωρήσει. Θα θέλαμε βεβαίως να βάλουμε και τα SDGs δηλαδή τις γενικευμένες προτιμήσεις, την εμπορική μας πολιτική, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το κάνουμε μέσω των εμπορικών διαπραγματεύσεων με, τρίτους, με τρίτες χώρες. Ο πρόεδρος μίλησε για την δέουσα επιμέλεια, η Κομισιόν μίλησε για την Πράσινη Συμφωνία και ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην διακυβέρνηση των εταιριών. Και ετοιμάζουμε και δύο μελέτες για την δέος επιμέλεια στην αλυσίδα ανεφοδιασμού. Η μελέτη αυτή θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες και για την... Ε, τον Απρίλιο του 2020 θα έχουμε τη μελέτη για την ε, ε, διακυβέρνηση των εταιριών, την εταιρική διακυβέρνηση. Θα επανέλθουμε λοιπόν για αυτά τα θέματα. Πολύ ωραία. Για το δεύτερο κύκλο έχω... 19 συνάδελφες ζητούν το και αυτό σημαίνει 1,5 λεπτό αυστηρά ο καθένας. Σύντομα και βρώμικα. Είμαι Ροντρίγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την παρέμβασή σα, τη σαφέστατη παρουσίασή σα. Θα επικεντρωθώ σε μία σειρά από ερωτήσεων. Μιλήσατε για συντονισμό ανάμεσα στην εμπορική πολιτική και τη βιομηχανική πολιτική. Τι συντονισμό εννοείτε ότι θα κάνετε Ποια θέματα θα ενισχυθούν για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας για τη γεωργία. Ως Επίτροπος γνωρίζετε πάρα πολύ τα, καλά τα προβλήματα του κλάδου. Πολλές από, τα, από τις ε, παρατηρήσεις και τα παράπονα που ακούμε είναι ότι οι τρίτες χώρες δεν σέβονται τα φυτοϊγειονομικά πρότυπα και ούτε έχουν περιβαλλοντικά πρότυπα. Εκείνες οι χώρε ενώ εμεί έχουμε και αυτό είναι πιο αποτελ... ε, σημαίνει το σύστημά μας είναι πιο αυστηρό. Ε, από την άλλη, συχνά κάποιε από αυτέ τι χώρε έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά μας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό το θέμα, για αυτή τη διαφορά δηλαδή αντιμετώπισης. Τώρα, για τους α, ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με ανησυχεί το γεγονός ότι καθυστερούμε να αναγνωρίσουμε μια κατάσταση που έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή, να μην καθυστερούμε τόσο δηλαδή. Κυρία Καβατσίνη. Ευχαριστώ, Επίτροπε, και χαίρομαι που είστε εδώ. Είναι καλή ευκαιρία να έχουμε διαρθρωμένο διάλογο Πρώτα απ' όλα να αντιδράσω σε κάποια από αυτά που είπατε. Πρώτα απ' όλα ε, βλέπουμε θετικά αυτό που έγινε αλλά χθε στη, στην Ολλανδία ήταν όντω πολύ μικρή διαφορά και καλό θα ήταν να δούμε με την Επιτροπή την κατεύθυνση της εμπορική πολιτικής. Είναι πολλοί πολίτες και η Βουλή στην Ολλανδία που είναι πολύ επικριτική κατά της συμφωνίας. Είναι πολύ εύκολο να λέτε ότι δεν έχει προβληθεί σωστά. Σίγουρα υπάρχει γι' αυτό ένα πρόβλημα, αλλά καλό να το συζητήσουμε. Και μετά για το κατά πόσο εφαρμόζονται τα κεφάλαια TST. Ε, εδώ δεν έχουμε ανωνυμία, πόσο μάλλον. Και είχαμε αποφασίσει ότι η καλή εφαρμογή των κεφαλαίων τεστ είναι πολύ σημαντική και ήταν ένα σαφέ μήνυμα προ εσά για να εφαρμοστεί από το Κοινοβούλιο. Και ε, το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό που λέτε, ότι το κλίμα θα είναι κεντρικό θέμα όλων των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Εννοείται ποιε μελλοντικέ εμπορικέ ε, μπορείτε να μας πείτε ποιες εμπορικές συμφωνίες εννοείται για το μέλλον. Κάποιες θα τις επαναπτυαγαδευτούμε ίσως, κάποιες δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρωθούν. Είναι πολλές αυτές που έχουν μείνει Είναι ας πούμε η συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία αυτές που υπόψη. Και το θέμα των φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα τα έθεσαν ε, και δύο τουλάχιστον συνάδελφοι. Υπήρξε αίτημα πληροφόρηση από την κοινωνία των πολιτών, ναι, ολοκληρώνω. Το οποίο ήταν πολύ ενισχυτικό, γιατί δείχνει ότι πολλά από αυτά που ε, λέτε, ε, ε, η Αυστραλία, ο Καναδά πιέζουν, πιέζουν να αλλάξουμε τα επίπεδα των επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων. Ε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι και στι συνομιλίε με τι υπόλοιπε δεν υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ραφαέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα Ολλανδικά. Επίτροπε, ευχαριστώ, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το απόγευμα. Ελπίζουμε να σας βλέπουμε πιο συχνά στο μέλλον στην, Διεθνή Επιτροπή, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, το μέλλον είναι αβέβαιο. Όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα, Υπάρχει σχετική υποστήριξη για τι εμπορικές μας συμφωνίες. συμφωνίε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα εάν ε, περάσουμε και σε άλλε συμφωνίες... Και εγώ αυτή την πρόκληση τη βρίσκω υπέροχη. Χθε ε, η κάτω βουλή των κάτω χωρών ε, εψήφισαν με μικρή διαφορά υπέρ τη συμφωνία και βάσει αυτή τη ε, πλειοψηφία μένουν αφιβολίες για το αν θα εγκρίνει και η Άνω Βουλή την συμφωνία. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι μέτρα θα μπορούσατε να αναλάβετε αν τα κράτη-μέλη καταψηφίσουν την κύρωση συμφωνία όπως η ΣΕΤΑ. Ε, τι ε, συνέπειες υπάρχουν για τις συμφωνίες αυτές καθεαυτές και υπό το φως όλων αυτών των εξελίξεων. Πώς βλέπετε το μέλλον της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Όπως είπα, είναι μια πραγματική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εάν θέλουμε να αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο το διεθνές εμπόριο ώστε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Και επίσης για το εμπόριο και το κλίμα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να είναι πραγματικά μια συνιστόσα των μελλοντικών εμπορικών μας συμφωνιών. Ε, πρόεδρε, ε, ευχαριστώ. Θα περάσω τώρα στα Ιταλικά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, Επίτροπε. Θέλω να επικεντρωθώ στις ΕΠΑ διότι είναι για, πολλά, για πολλούς ενδιαφερομένους ένα σοβαρό πρόβλημα και πρέπει κάπως να δούμε τι θα κάνουμε με την εμπορική τους επιθετικότητα, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε. Πώς θα επιδιώξουμε όμως αυτό το στόχο, όπως ε, πολλοί ενδιαφερομένοι ανησυχούμε για την επιστηστική ασφάλεια λόγω χάρη. Γι' αυτό πολύ γρήγορα κάποιες ερωτήσεις. Για τα φυτοφάρμακα έχει γίνει πολλή κουβέντα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν πέραν των φυτοφαρμάκων, υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε αμοιβαία αναγνώριση για τα προϊόντα που έχουν να κάνουν και με την επεξεργασία κρέατος. Η δεύτερη ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εντολή τη για να γίνονται κάποιε αξιολογήσει συμβατότητα και να αλλάξουν κάποια υγειονομικά πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι οι ΙΠΑ τα θεωρούν μη δεσμολογικού φραγμού. Και το τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναξιολογεί με την ΕΦΣΑ τη δυνατότητα να εγκριθούν κάποια γάματα φόμικρων. Ε, και η ερώτησή μου είναι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να αλλάξει ε, για κάποια αμερικανικά προϊόντα ε, τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Ευχαριστούμε κύριο Μπορέλ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Είπατε, Επιτροπέ, ότι το εμπόριο είναι ένα εργαλείο για να ε, προωθήσουμε, να καλλιεργήσουμε έναν ε, κόσμο σε ευμάρεια. Όμως είστε σίγουρος, γιατί το πρωί κοιτάζοντα ε, τον προπολογισμό της Επιτροπής και αυτά που προτείνονται, είδαμε ότι με την αύξηση των ελευθέρων συναλλαγών ε, αυξάνει το όγκο των συναλλαγών, αλλά όχι ε, τα εργασιακά δικαιώματα ή η προστασία του περιβάλλοντο. Δεν υπήρχαν τέτοιε ρήτρε ε, στι παρελθούσε συμφωνίε, δεν θα υπάρξουν στι μελλοντικέ. Πώ θα προωθήσουμε την Πράσινη Συμφωνία και θα διπλωματευτούμε με την Ινδονησία που είναι πρωταθλητή τη αποψήλωση παγκοσμίω. Πώ ε, θα μιλάμε για την βιωσιμότητα και μετά για την Αυστραλία με τι χειρότερε επιδόσει για την προστασία του περιβάλλοντο που είναι πιο μακριά από όλε από την Ευρώπη, θα εντατικοποιήσουμε τι εμπορικέ σχέσει. Εκεί οι κουμπέ δεξιού του άνθρακα είναι καταστροφικέ. Εδώ λοιπόν, εντάξει, τα λέτε θετικά, αλλά ε, μα τα λέτε πολύ καθησυχαστικά. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Ε, δεν πάνε καλά. Γιατί θέλω να κλείσουμε τι ΗΠΑ σήμερα. Έχουμε με μια πολιτική εξόχως επιθετική. Ε, εδώ πραγματικά μιλάμε για την εξοδαφικότητα του Αμερικανικού δικαίου, για επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείε που έχουν εμπορικέ σχέσεις με το Ιράν, ε, εταιρείε που μπορεί να βοηθήσουν να ε, ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα, ένα έργο που το λέμε Nord Stream 2. Δεν είναι στη ΣΥΠΑ, είναι στην Ευρώπη αυτά. Και τι κάνουμε σήμερα, συζητάμε για ένα μίνι TTIP, την παλιά συμφωνία που είχαμε πετάξει έξω μεγαλοπρεπώς, κλωτσιδών και τελικά θέλουμε να τη βάλουμε από το παραθυράκι. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη κάπως πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ευχαριστούμε κυρία Γκριμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για σας. Η πρώτη αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανακοινώσατε ε, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τη συμφωνία με την Καμπότζη και είπε ότι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ε, είναι ότι είναι διαπραγμάτευτα και αναπαλωτρίωτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά τις, τα βήματα πρόοδου όμω, είναι πολύ ε, κρίσιμη και ανησυχητική κατάσταση στην πράξη. Συμφωνούμε λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί σα, όμω πρόσφατα συζητήσαμε και μάλιστα εντόνω για το Βιετνάμ. Για τα μέτρα λοιπόν που σκέφτεστε να θετήσετε, τι κριτήρια ανάλυσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σκέφτεστε να αποκρινέτε, τι θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κριτήριο στις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες και στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, για να έχουμε και μια γραμμή ε, συνοχής μεταξύ των θέσεων των κρατών μελών και αυτών που υιοθετούν και όργανα όπως ε, η ΕΕΔ, και η οποία έχει πολλά παρεδόσει με το Βιετνάμ, λόγου χάρη. Και μετά για τον μηχανισμό μηδενική ανοχή, για την παιδική εργασία, λόγου χάρη. Τι ακριβώ θα κάνετε. Και να επαναλάβω και εγώ την ερώτηση για αυτά που αφορούν το ε, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το φύλλο και ε, ε, πώς θα εντάξει αυτή τη ε, διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μια η Πράσινη Συμφωνία, από την άλλη ε, το σύστημα επίλυσης διαφορών, πώς θα προστατεύουμε τις ε, βιώσιμες επενδύσει. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Σχετικά με τις συνεχιζόμενες δια, δια, ε, διαπραγματεύσεις με τον Ηνωμένο και σε σχέση με την Βόρεια Ορλανδία υπάρχει ένα πρωτόκολλο που την τοποθετεί σε μια ανευπροηγουμένου θέση σε σχέση με τις σχέσεις με τρίτες χώρες. Πρώτο ερώτημα είναι, αν έχει ληφθεί υπόψη το αν μπορεί να επιλε... ε, ε να επωφεληθεί από τις μελλοντικέ εμπορικές συμφωνίες ε, η Βόρεια Ιρλανδία και επίσης στον τομέα των ε, ε, υπηρεσιών όπως και στα αγαθά. Επίσης έχει, έχουν ληφθεί υπόψη η σωστή εκπροσώπηση των συμφερόντων της Βόρειας Ιρλανδίας γιατί όπως είπαμε υπάρχει σε μοναδική, είναι σε μοναδική θέση. Ας πούμε η μερική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το πρωτόκολλο, για, τα, για την ενιαία αγορά ηλεκτρισμού στην νήσο της Ιρλανδίας. Επίσης, αν δεν έχουν όλα τα μέλη ε, κυρώσει ε, την, μια μελλοντική συμφωνία μέχρι 31η 12 του, του ε, 20, τι προτείνετε για, την, ε, για τα προβλήματα στο εμπόριο μέχρι τότε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Μία για τι διαπραγματεύσει, εμπορικέ διαπραγματεύσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακούμε πολλά μηνύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το τι περιμένουν να επιτύχουν από την ε, ε, Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου. Περιμένουν ότι θα έχουν ε, τη δυνατότητα να θεσπίσουν δικούς τους νόμους. Τι θα συμβεί αν αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο να μην τηρήσει τους κανόνες για τον δίκαιο και ανοιχτό ανταγωνισμό. Τι σημαίνει ότι ε, δεν θα γίνονται αποδεκτές οι βρετανικές επιχειρήσεις. Φυσικά θα θέλαμε να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά ποια θα είναι η θέση μας επ' αυτού σε σχέση με μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλες ε, ρεαλιστικές συμφωνίες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, όπως με τον Καναδά και την Αυστραλία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τις ΗΠΑ. Στην Ολλανδία λέμε ότι όταν ε, τσακώνονται δύο σκυλιά για το ένα κόκαλο υπάρχει ένα τρίτο που το αρπάζει και φεύγει και διερωτώ με ποιος θα είναι ο τρίτος στην περίπτωση αυτή. Ε, εδώ που χαίρομαι που εξακολουθούμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο με τις Ηνωμένε Πολιτείε και υπάρχει κάποια κίνηση στον τομέα της αγοράς των ε, δημοσίων συμβάσεων. Από αμερικανικής πλευράς εννοώ. Ευχαριστώ. Κύριο Σάρτη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προκάτοχό μου για την προλαλήσασα, γιατί ρώτησε ακριβώς αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω. Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, ε, με το μέλλον των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, άρα το ξεπερνάω αυτό και ως εκ τούτου μου μένει μόνο μία ερώτηση για την Κίνα. Παρακολούθησα τον κύριο Μπορέλ πέρσι στην διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου. Εκεί είπε ότι όλο και περισσότερο υπάρχει ένας διπολισμός στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας και ότι θα πρέπει η Ευρώπη να προσέξει να μην παγιδευτεί ανάμεσα στα δύο, αυτούς δύο αυτούς πόλους. Πώς ε, εντάσσεται αυτό ε, στην ε, εμπορική στρατηγική σας για τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα που θα και βεβαίως υπό το φως της τρέχουσας κρίσης με τον νέο ιό που, γιατί και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη στρατηγική του στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έδωσε καρπούς. Πολλές ανησυχίες των γεωργών, των βιομηχάνων ε, που παράγουν τρόφιμα στην Ευρώπη είχαν, ήταν τρομοκρατημένοι πριν λίγες μέρες. Τουλάχιστον ε, τις τελευταίες μέρες μας φτάσαν ειδήσει ότι δεν αλλάζει τίποτα, τουλάχιστον προς το παρόν. Ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα στη στρατηγική με τον ΠΟΕ και να λυθεί και το πρόβλημα με τους δασμούς των Αμερικανών. Η κατεξιοδότηση πράξη για την Καμπότζη λόγω της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στον κατάλογο προϊόντων δεν αναφέρεται το ριζί. Αυτό μας ανησυχεί, γιατί όπως ξέρετε η ρήτρα διασφάλισης που ισχύει λίγη τον Ιανουάριο του 2021. Θα ήταν ίσως χρήσιμο λοιπόν σε αυτή την ε, κατεξιοδότηση πράξη να γίνει μία δήλωση της Κομισιόν ότι αν οι συνθήκες αγοράς συνεχιστούν και παραμείνουν ίδιες με σήμερα, η Κομισιόν θα συνεχίσει με αυτή τη ρήτρα διασφάλισης. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να εξηγήσουμε γιατί δεν υπάρχει το ρύζι σε αυτή την λίστα προϊόντων, σε αυτόν τον κατάλογο προϊόντων. Ευχαριστώ. Βίνκλερ, uh, ευχαριστώ Πρόεδρε ε, και πάλι είναι χαρά, μου, χαρά μας να σας ακούμε και να έχουμε ευκαιρία για διάλογο. Ερωτήσεις. Ε, για την Κίνα. Το σχόλιο μου θα ήταν σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά ε, την προοπτική των εμπορικών μας σχέσεων, σας ρώτησε ο κύριος ε, Σόλτς τι θα γίνει με τη λειψία. Το ΕΛΚ θα έλεγε ε, για το χρονοδιάγραμμα, για την ποιότητα. Αλλά δεν είναι μόνο η προθεσμία, είναι το περιεχόμενο που μας νοιάζει. Επίσης, σε αυτή τη φάση έχουμε συμφωνία που διαβλέπουμε, είπα, Κίνας. Ε, Χθε στην Επιτροπή Γεωργίας είδαμε πώς μπορεί να επηρεάσει επηρεάσει μια τέτοια συμφωνία τη δική μας της, ε, με την Κίνα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Και Εάν υπάρχει συμφωνία επακίνα, τι θα γίνει με τι δικέ μα τι γεωγραφικέ ενδείξει. Και η δεύτερη ερώτηση, αναφέρατε τον ΠΟΕ και την ανανέωση των ε, μηχανισμών διευθέτηση διαφορών. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έχουμε 16 κρατημέλη που ενδιαφέρονται και το συζητήσατε ενδεχομένω με Κινέζου συνομιλητέ. Η Κίνα θα ενδιαφερόταν να συμμετάσχει σε αυτή την ενδιάμεση, την προσωρινή συμφωνία. Ο κύριος Χαβιέρ Μορένο. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, χαίρομαι που είναι εδώ ο Επίτροπος και ακούσαμε ένα καλό νέο. Έχω, είμαι, έχω το ρόλο του εισηγητή για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Η Ολλανδική κυβέρνηση, η Ολλανδική Βουλή, συγγνώμη, επιτέλους είπε ναι. Δεν ξέρω ποια είναι τα επόμενα βήματα, που είναι σημαντικά όμως. Ε, και αυτοί που μοιάζουν πιο Ευρωπαίοι εκτός Ευρώπης είναι οι Καναδοί. Ε, η προσωρινή εφαρμογή έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα και για τους μεν και για τους δε. Ξεκινήσαμε με διάφορες αρχές, σε διάφορα επίπεδα του Καναδά ε, και όλοι μου είπαν ότι ήταν θετικές οι επιπτώσεις της προσωρινής εφαρμογής. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, τόσο ώστε αυτή η προσωρινή ε, συμφωνία να γίνει οριστική συμφωνία. Ο νόμος Helms-Barton δημιουργεί ανησυχίες όλο και περισσότερο στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Κούβα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thanks, Chair. Muchas gracias, κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, για τη διαφάνεια και τα πρότυπα και σε σχέση με τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ. Ανησυχεί βαθιά πολλού πολίτε ανά την Ευρώπη, ιδίω για το γεωργικό τομέα στην Ιρλανδία, α πούμε. Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Και ακούσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώνεται τι γενικέ διατάξει την περασμένη εβδομάδα. Με αυτά από τα κεφάλαια για τι δημόσιε προμήθειε. Πώ πάει εκεί το πράγμα, η Γενική Διεύθυνση Trade, η ΕΕΔ για το πολιτικό σκέλο συνεχίζει να διαμορφωτεύεται και άλλα κεφάλαια για τη Συμφωνία Μερκοσούρ, αφού πριν από μερικού μήνε ακούσαμε ότι έχουν διαθετηθεί. Ε, κάνετε τώρα το νομικό νοικοκύρεμα. Ε, και αν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει, ποια είναι τα τμήματα που σα ενδιαφέρουν ε, σε αυτή τη φάση. Και μετά για τα σχόλιά σα σε σχέση με, την, ε, με τι ΗΠΑ. Σίγουρα, να μην, διαβάζουμε, να μην πιστεύουμε ότι διαβάζουμε στι εφημερίδε. Εγώ θα το πω πρώτοι αυτό. Αλλά πολλά έχουν υποθεί και καλό θα ήταν να μας καθησυχάσετε λίγο παραπάνω, διότι έγινε πολλή κουβέντα για το πώς είπα, ε, θα επιτρέψουν ε, στις αγορές μας προϊόντα με, με χλωρίνη και ένα σωρό άλλα προϊόντα και κάποια κάποια άλλα που ως τώρα δεν ε, είχαν πρόσβαση. Τι θα κάνετε λοιπόν με τα πρότυπα ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά, γιατί και εδώ υπάρχει θέμα δημόσιων προμηθειών. Και μετά, όχι εντάξει, ολοκλήρωσα. Ο κ. Χάνσεν, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να παραμείνω στο 1,5 λεπτό. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, που είστε εδώ. Η πρώτη με ερώτηση είναι για την διμερή ε, συνθήκη, συμφωνία με την Ταϊβάν. Πώς σκοπεύουμε να το διαρθρώσουμε με τις διαπραγματεύσεις με την Κίνα. Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι ότι ακούμε να υπάρχει κάποια κίνηση για την ε, Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων στο Συμβούλιο οι διαπραγματεύσεις αυτές όντως προχωρούν ή ήταν απλώς ε, δουλειά καλοπιστική αυτή που έγινε. Και μετά ξέρετε ότι είμαι συγκεκριτής αυτή τη επιτροπή για τις μελλοντικές σχέσεις την εξέλιξη μάλλον και το τι μορφή συμφωνία θα έχουμε, ελεύθερων συναλλαγών ενδεχομένω, με το Μενό Βασίλειο. Την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλε ακούσαμε τον κύριο Τζόνσον σε μια ομιλία του να λέει ότι έχει τη δική του άποψη για το θέμα αυτό. Εσεί ίσω, επειδή δεν είστε Βρετανό και είστε Ιρλανδό, να έχετε διαφορετική άποψη για αυτά τα πράγματα και να μπορείτε κάτι να μα πείτε. Η διαδικασία εδώ πάντω, και επειδή δεν ε, συμμετέχουν απευθεία όλοι οι συνάδελφοι, μπορείτε να μα πείτε ποια είναι τα βασικά θέματα που θα μα απασχολήσουν, οι προτεραιότητε και το χρονοδιάγραμμα. Ακούμε ότι το Συμβούλιο θέλει να διευρύνει το πεδίο των δημοτεύσεων. Τι ακριβώ θα κάνετε εκεί. Ευχαριστώ, κύριε Κάνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τις μεγάλες απειλές του διεθνούς εμπορίου. Εσωτερικές και εξωτερικές. Τρεις ερωτήσεις για τις εξωτερικές. Μονομέρια, διπλωματία και δασμή της κυβέρνησης Τραμπ. Τι θα κάνει η Κομισιόν μπροστά στις απειλές Τραμπ. Ε, απέναντι στις χώρες που εφαρμόζουν ε, ε αυτό το φόρο κυρίως ε, ε, για τις τεχνολογικές εταιρείες γιατί φοβούνται τους δασμούς ε, τον των ΗΠΑ. Τώρα, εσωτερικές απειλές. Ο Επίτροπος μίλαγε για ισορροπία. Κοιτάξτε, τι θα γίνει για τους... Ε, για για, γιατί να μην μιλάμε καλύτερα για ισορροπημένο παιχνίδι. Ε, έχουμε 11 παίχτες, ας πούμε, στο, στο ποδόσφαιρο. Ε, είναι δύσκολο να παίζουμε διαφορετικού κανόνε. Υπάρχουν, α πούμε, 11 παίκτε στην ε, ομάδα, οι 10 παίζουν του κανόνε και ο ένα παίζει με τα χέρια, α Τι θα γίνει, είναι κουραστικό για του υπόλοιπου. Επίσης, ε, έχουμε το Συμφωνία του Παρισιού, ε, το Green Deal ε, που μπαίνουν στα εμπορικά θέματα. Πώς θα επηρεάσει η Green Deal, τι νέε εμπορικέ συμφωνίες, η αναδιαπραγμάτευση, πώς θα επηρεάσει την αναδιαπραγμάτευση των ισχυουσών συμφωνιών. Επίτροπε, αν θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου η μέτρηση το άνθρακα θα θεωρείται φόρος, πρέπει να την απομακρύνετε από την Γενική Διεύθυνση Τάξουτ. Επίσης, ήθελα να σας ρωτήσω για την ε, συμφωνία της πρώτης φάσης και η, πρώτη σας αντίδραση ήταν σχετικά αρνητική. Εκ των υστέρων όμως πέρασε λίγος καιρός και ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η Κομισιόν ε, εξετάζει ε, τις ε, συνέπειες Επίσης, αν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει νομικά. Ευχαριστώ. Κύριε, κύριε ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτον, ευχαριστώ τον κύριο Χόγκαν, τον οποίο πρέπει να επανέσουμε για τα διαφανή του σχόλια. Έχουμε ένα διαφανή επίτροπο, οι Ιρλανδοί συνάδελφοι ρώτησαν για την Ιρλανδία και τον Brexit. Εγώ θα τα αφήσω αυτά και θα ε, ασχοληθώ με τα θέματα του οποίου είμαι ε, μόνιμος συζητητής. Η, λίγη το 23 η παρούσα συμφωνία για τη σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Ε, πώς βλέπετε τα πράγματα, κυρίως σε σχέση με το κατά τους οποίους, το, τους οποίους ψήφισε πέρυσι το Κοινοβούλιο για την διαφοροποίηση, ε, την βελτίωση των ε, περιβαλλοντικών προτύπων και την ενισχυμένη εποπτεία. Και επίσης ε, σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες θα ήθελα το Κοινοβούλιο, να, χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ήταν τόσο πολύ υπέρ τη συμφωνία με το Βιετνάμ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε και συμφωνία με, με την Ινδονησία και οποιαδήποτε προσπάθεια Υπάρχουν ειδήσει για το τι θα γίνει με τη Μαλαισία τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το ταχαίως ε, αναπτυσσόμενο κομμάτι του κόσμου. Ε, ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κ. Σούτσι. Θα, θα μιλήσω Ιταλικά. Για τη συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ, τι ε, προθέσεις έχετε, διότι έχει επιβεβαιωθεί η διάθεση κάποιου τους μέλους μιας κυβέρνησης να μην υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε αυτό τον ε, σκόπελο. Ε, ε, νομίζω είναι θεμητή ερώτηση, διότι είναι η πολλαπλή ε, απόπειρα εμπορική συμφωνίας την οποία κάποιος μπλοκάρει και μιλάμε για μηχανικά προϊόντα στα γεωργικά, στη γεωργική μας παραγωγή. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έχει συνέπειες και για τους καταναλωτές. Έχετε σκοπό να διαιρέσετε την συμφωνία σε ε, δύο σκέλη εμπόριο επενδύσεις για να ξεπεράσετε αυτό το σκόπελο των κατομελών. Συμφωνία ΙΠΑ Κίνας. Έχετε την ε, πρόθεση να προχωρήσετε σε λεπτομερέστερη εξέταση για να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ευρωπαϊκές εισαγωγές προς την Κίνα και για τον ΠΟΕ. Έχετε την πρόθεση να θέσετε το ερώτημα διότι η Κίνα έχει δεσμευτεί για την ε, ε, απόκτηση και την αποδοχή αμερικανικών προϊόντων. Οπότε όλα αυτά είναι συμβατά ε, με τους κανόνες του ΠΟΕ που τόσο πολύ θέλετε να προασπιστείτε ή όχι. Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εντάσει στον ΠΟΕ. Τι δράση σκοπεύετε να αναλάβετε στη Γενέβη προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την ε, επίσκεψη και την αντίδρασή σας. Θα ήθελα να επανέλθω ε, σε θέματα όπως ας πούμε η διαφωνία του Airbus, της Airbus Συμφωνώ με το, την ανησυχία του κόσμου της αεροπλοείας. Ε, είναι καλό να υπάρχει επι, ε, επικοδομικός διάλογος, αλλά μερικοί έχουν, κάνουν τους κοφούς. Αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τη, τα ε, συμφέροντά μας. Υπολογίζουμε σε εσά Όσον αφορά τον ΠΟΕ ευρύτερα, ε, αναφερθήκατε στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα όμω περισσότερες συγκεκριμένες διευκρινήσει για τις προσδοκίε και τους συγκεκριμένους ε, στόχους σα ε, εν ώψη της Υπουργική του Ιουνίου και επίσης σε σχέση με την Κίνα, είπαν και οι συνάδελφοι, είναι πολύ καλή είδηση ότι έχουμε εν ώψη συμφωνία Κίνας, με τις διατάξεις σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία και τα ε, εμπορικά σήματα, ποιες θα υλοποιηθούν και οι γεωγραφικές ενδείξεις στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, βλέπετε ότι η Επιτροπή γνωρίζει πολλά πράγματα στον τομέα της βιομηχανίας. Ε, έχουμε πολλές ερωτήσεις και ξεκάθαρες θέσεις. Και τώρα έχετε το θαυμαστό καθήκον να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά εντός δεκαλέπτου. Είμαι, είμαστε και ευέλικτοι όμως, αν θέλετε πιο πολύ χρόνο. Έχω γίνει πολύ ε, σε αυτά τα θέματα τα τελευταία χρόνια. Ε, Ο Επίτροπο Μπρετών είναι υπεύθυνο για τη βιομηχανική πολιτική και αυτή τη στιγμή συζητάμε και θα δούμε τι θα έχουμε κάνει ω τότε μέχρι να ξεκινήσουμε τη βιομηχανική μα πολιτική το εμπόριο είναι σοβαρό σκέλος και πρέπει να συνδυαστεί με τη βιωσιμότητα. Η Πράσινη πάντω συμφωνία είναι ευκαιρία διότι έχουμε υπάρξει πρωταγωνιστές ό,τι αφορά την ε, βιωσιμότητα ε, και την ε, δημιουργία, την παροχή τεχνολογικών λύσεων για να μπορούν οι εταιρείε να πουλάνε στους πολίτε ανά τον κόσμο με τα σωστά πρότυπα για την βιωσιμότητα στα προϊόντα μα στη μηχανοποίηση τη γεωργία. Τα γνωρίζω πολύ καλά λοιπόν. Εγώ έχω επίγνωση τη κατεύθυνση στην οποία οδεύουμε. Και βεβαίω υπάρχουν ανησυχίε όπω την αμοιβαιότητα, τα πρότυπα. Έχουμε δαπανίσει πολύ χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια προσπαθώντα να ξεπεράσουμε του μη δεσμολογικού φραγμού και να έχουμε ισότιμου ε, όρου ανταγωνισμού για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε σε σχέση με άλλε. Κάποιε φορέ, οι φραγμοί δεν είναι για σκοπού κοινή λογική εκεί, είναι για πολιτικού λόγου. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάμε να μην έρχονται προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνατών που να μην ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι πολλά τα κρατημέλη που περνάνε χρόνο και δαπανάνε πόρου για τι επιθεωρήσει και του έλεγχου για να μην συμβεί αυτό. Για να έχουμε ψηλά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να τα προστατεύουμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνονται αυτά σωστά. Ε, για τους ε, φραγμούς ε, στην αγορά μας και το τι συμβαίνει με, το, με τα μέτρα SPS. Αυτά πολλές φορές υπάρχουν για πολιτικούς λόγους. Δεν είναι θέματα μόνο δημόσιας υγείας ή υγιεινής. Δεν συμφωνώ με την αποτίμησή σας για την συμφωνία ΣΕΤΑ και ε, θα το περιμένατε. Ε, Εσεί είσαστε εναντίον τη ΣΕΤΑ από ό,τι φαίνεται, ενώ εγώ την θέλω τη συμφωνία αυτή. Ε, και εν τέλει είναι θετικό το αποτέλεσμα. Η Ολλανδία τελικά υπερψήφισε τη συμφωνία. Εγώ είμαι ικανοποιημένο με αυτή την έκβαση. Είναι θετικό αυτό που συνέβη. Τώρα, εάν όντω ε, ε, περάσει η συμφωνία, νομίζω ότι ο κόσμο χάρηκε που μπόρεσε να αντιμετωπίσει και την παραπληροφόρηση που δεχόμασταν από την προπαγάνδα κάποιων άλλων πηγών. Τώρα, για την TST και την δυνατότητα να εφαρμοστούν τα κεφάλαια αυτά στην πράξη, η κάθε συμφωνία προτείνει τι δομέ που πρέπει να δημιουργηθούν, τι μορφέ διαλόγου, σε απουσία αυτών τι κυρώσει. Εάν χρειαστεί, λοιπόν, θα κοιτάξουμε να έχουμε ανάλογε διευθετήσει για να διασφαλίσουμε την πραγματική εφαρμογή των διευθετήσεων action ε, Βεβαίω κάποια δεν προχωρούν αρκετά αγοργά ε, όπω θα θέλαμε. Έχουμε όμω επιμέρου διαδικασίε για να τα ελέγχουμε αυτά και εν τέλει, ε, όπως στην περίπτωση τη νότια Κορέα, είναι ένα τέλειο παράδειγμα το τι κάνουμε στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα για να, για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αναθεώρηση των συμφωνιών που προβλέπουμε. Βάσει των εμπειριών που έχουμε τώρα, η Καμπότζη είναι ένα άλλο παράδειγμα, θα επανέλθω σε αυτό σε μισό λεπτό. Όμω, Εάν είμαστε σοβαροί ότι θέλουμε συμφωνίε, ευθύ εξ αρχή, δεν μπορούμε να μην πάμε ως εκεί. Και δεν μπορούμε και να πάμε και παραπέρα για την ώρα. Έχουμε πετύχει πολλά με τη Συμφωνία Μερκοσούρ, κατά την άποψή μου, η αρχή τη προφύλαξη. Η Συμφωνία των Παρισίων. Η Βραζιλία δεν ήθελε καν να πάει σε την κατεύθυνση αυτή. Ουδέποτε. Όμω, οι συνεισφορές ε, DNDC που περιμένουμε από τη Βραζιλία ελπίζουμε ε, να υπάρξουν. Ιδάλλως αναστέλλεται πλήρως η συμφωνία. Αυτό είναι η άλλη επιλογή. Δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά μπορεί να φτάσουμε και σε αυτή την κατάσταση. Δεν είμαστε όμως εκεί ακόμα για τις μελλοντικές συμφωνίες. Το λέω μόνο αν έχουμε εντολή. Μόνο αν πάρουμε εντολή για μελλοντικές συμφωνίες. Ήταν υποθετικά όλα αυτά. Ξέρετε τις απαντήσεις, τις ξέρετε πριν τις ρωτήσετε είναι σαφέ την ανακοίνωσή μα ε, για όλε τι μελλοντικέ ε, σφαιρικέ και ει βάθο συμφωνίε μα για το εμπόριο. Το θέμα της Συμφωνίας των Παρισίων, το σκέλος αυτό θα πρέπει να έχει μπει στο κείμενο, ε, να έχει ενσωματωθεί δεν μπορείτε όμω να περιμένετε να αλλάξουν οι κανόνε ε, χωρί διαπραγμάτευση. Ε, αν έχουμε κάποια εντολή. Μελλοντικά. Βεβαίω η Συμφωνία των Παρισίων θα είναι ένα συστατικό στοιχείο τη κάθε συμφωνία. Για το τωρινό επίπεδο, ναι, παρακαλώ. Δεν ήταν σαφέ. Ναι, ναι, σαφέ ήταν. Όμω δεν έχουν μείνει συμφωνίε πλέον στον κόσμο. Δεν έχουμε πια συμφωνίε στον κόσμο. Εάν πάνε έτσι τα πράγματα. Ε, εγώ σα λέω την πραγματική μα στάση. Τώρα είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε. Ε, το ξέρω ότι διαφωνείτε. Αλλά οι μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε, οι μελλοντικέ σφαιρικέ και ει βάθο εμπορικέ συμφωνίε θα συμπεριλαμβάνουν ω αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο τη Συμφωνία των Παρισίων. Αυτό είναι το γεγονό. Τώρα, τα τωρινά όρια για τα φυτοφάρμακα και για τα προϊόντα των ΗΠΑ δεν θα αλλάξουν αυτή τη στιγμή, δεν θα μειωθούν προ τα κάτω. Και για, παθογεν, για του παθογενεί παράγοντε και για τα MRL, ε, τα κατάλοιπα, το λέω για να μην ανησυχείτε δείτε, δεν αλλάζουμε τώρα τους κανονισμούς, ούτε θα κάνουμε καμιά τέτοια συμφωνία στο περιθώριο. Κυρία Ραφαέλα, η θέση σας για το εμπόριο το εμπόριο είναι ευθύνη όλων μα εφόσον ε, εργαζόμαστε ω ε, συνεργάτε. Η δικιά σα θέση στο εμπόριο στην Ολλανδία είναι κάτι που να προωθήσετε. Αν είστε υπέρ του εμπορίου, προωθήστε αυτήν την έννοια. Ε, να το δει και ο κόσμο. Εάν έχετε ανησυχίε, εκφράστε τι. Όμω η ευθύνη είναι όλων μα. Πρέπει να πούμε ποια είναι τα ωφέλη του εμπορίου και να το καταλάβει ο κόσμο. Εάν δεν το πετύχουμε αυτό και αν υπάρξουν προβλήματα μάλλον και αυτά πρέπει να τα εντοπίσουμε. Ο καθένα πρέπει να αναλάβει τι δικέ του ευθύνε και αναλαμβάνουμε όταν ψηφίζουμε είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό είτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν σκεφτόμαστε το εμπόριο, να σκεφτούμε τι εμπορικέ συμφωνίε διεθνώ και γενικότερα. Να το σκεφτείτε και στην Ολλανδία. Υπήρξε πολύ παραπληροφόρηση στην Ολλανδία για τα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι σε κάποιε περιπτώσει πέτυχε το σκοπό, του, ε, το σκοπό τη η παραπληροφόρηση τι θα γινόταν αν δεν είχαμε υπερψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Εγώ τώρα δεν θέλω να προβλέψω την κατάσταση, αλλά το Συμβούλιο είναι αυτό που τελικά θα αποφασίσει. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί που θα χρειαστεί να αποφασίσει το Συμβούλιο. Τώρα για το φύλλο, τη διάσταση του φύλλου στο εμπόριο. Όπω γνωρίζετε και το είπα και στι ακροάσει μου όταν είχατε ρωτήσει την ίδια ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική κοιτάζει να προωθήσει και του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη για την ισότητα των φύλων. Και προσφάτω ε, στι εμπορικέ μα συμφωνίε, στι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών, διαπραγματευτήκαμε μέσω του εμπορίου κεφάλαια για την ισότητα των φύλων. Οι διατάξει για το φύλλο ε, στι συμφωνίε αυτέ συμπεριλαμβάνονται ξεκάθαρα. Μπορείτε να τι κοιτάξετε ε, και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Η ποιότητα των όσων έχουμε πετύχει είναι κάτι που θα το καθορίσετε εσεί με τη δουλειά σα βεβαίω στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ε, Όμω είναι ε, προφανώ επιτάπητο ε, για τι συμφωνίε αυτέ. Ε, Πολλέ ερωτήσει τέθηκαν για τις σχέσεις μα με τη ΣΥΠΑ. Να το πω περιληπτικά ίσω και να απαντήσω έτσι σε όλους ταυτόχρονα. Για όσου ρώτησαν τι θα γίνει με τη ΣΥΠΑ και την Κίνα. Ε, για τις ΕΠΑ Λέτε να του ηρεμήσουμε κάνω ό,τι μπορώ. Το είδατε το πιο πρόσφατο παράδειγμα την Παρασκευή. Υπήρξε μια σχετική καλή θέληση. Θέλουν να μιλήσουν για πρώτη φορά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Αναστήλαμε την πρόβλεψη δασμών. Αφήσαμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία ανοιχτό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το εκμεταλλευτούμε. Θα το ξέρουμε σε 30 μέρες αλλά δεν θα μειώσουμε τα πρότυπα, δεν θα μειώσουμε τα, τις οριακές τιμές των φυτοφαρμάκων, των χημικών ουσιών, δεν θα πληγούν τα τρόφιμα και η παραγωγή τους. Ε, πραγματικά θέλω να διασκεδάσω όλες τις ανησυχίες που έχετε από τις φήμες που ακούστηκαν. Ε, έτσι κι αλλιώ. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ σε σχέση με τις εντολές που υπάρχουν, αυτές που μας έχετε αναθέσει εσείς για το εμπόριο και εκτός ε, των δημοτεύσεων εδώ. Ξέρετε την δήλωση του Ιουλίου Γιόνκερ Τραμπ. Ε, πολλά πρέπει, μπορούν να γίνουν εδώ. Η γεωργία ε, δεν περιλαμβάνεται, αλλά δεν πήραμε τις δημόσιες προμήθειες ας πούμε. Αυτό τώρα κοιτάζουμε να φέρουμε επιτάπητος. Εκεί είναι η διακριστήνδα και η παρανόηση κάποιες φορές. Κοιτάζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν συμφωνούμε πάντως με τον κύριο Μανουέλ. Ε, δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι το TTIP το παραθυράκι. Ήταν πολύ σφαιρική η συμφωνία η Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γίνεται τώρα. Για την Ινδονησία. Συνήντησα τον Υπουργό Εξωτερικών χθε και του κατέστησα σαφέ ότι αν δεν λύσουμε τα ζητήματα βιωσιμότητα και το φινικέλαιο δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ήμουν τελείω κάθετο. και το κατάλαβε. Υπάρχει ομάδα εργασία που προσπαθεί να καθορίσει τι θα γίνει με την Ινδονησία, τη Μαλαισία και άλλε τέτοιε χώρε και πώ θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του φινικέλαιο. Δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα για του όρου αναφορά. Ελπίζω να προχωρήσουν και να βρούμε του όρου αναφορά τι επόμενε μέρε για να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ξεπεράσουμε την ανατάραξη ε, όλη αυτή αλλά δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Ενδονησία ούτε θα ξανανοίξουν οι διαπραγματεύσει με τη Μαλαισία εφόσον δεν λυθεί το θέμα αυτό. Γι' αυτό σα διαβεβαιώ. Ε, νομίζω ο κύριο Μανουέλ με ρώτησε για την Αυστραλία ε, και το τι γίνεται με τα κεφάλαια ευαισθημότητα εκεί. Μα δεν θα υπάρξει συμφωνία με την Αυστραλία. Και ε, για το κεφάλαιο αυτό, εάν δεν φτάσουμε στον επίπεδο των φιλοδοξιών που έχουμε, όπω απαιτεί η εντολή μα, δεν θα προχωρήσουμε. Δεν θα το φέρουμε για ψηφοφορία στο ε, Ευρωκοινοβούλιο ή ούτε θα το παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο. Ψηφοφορία ε, τι να ψηφοφορήσουμε, τι να ψηφίσουμε αν ξέρουμε ότι ούτω ή άλλω θα ε, απορριφθεί. Καμιά φορά ο κόσμο δεν το καταλαβαίνει. Για την Καμπότζη. Για την Καμπότζη, κύριε Ντικάστρο και άλλοι που το είπατε, είναι πολύ απλό. Ε, χρειάζεται να δούμε τι θα γίνει με την κυβέρνηση της ε, Καμπότζης και την αντιπολίτευση. Εκεί πρέπει να αναλυφθεί η δράση. Πρέπει ε, να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία που έχουμε με την Καμπότζη. Και είναι αρκετή ε, βάση για να ξεκινήσει μια διαδικασία και να αποσυρθούμε από τη συμφωνία. Έχουμε έντονη δράση κατά της Καμπότζας προς στιγμή όμως. Ε, στις 22 Αυγούστου νομίζω είχαν ολοκληρωθεί κατά εξοδότηση πράξη. οπότε αν όλα πάνε καλά η Καμπότζη θα ανακαλέσει τις αποφάσεις της και θα κοιτάξει να ευθυγραμμιστεί με αυτά που περιμένουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχετικές πρακτικές και αυτά που περιμένουμε θα περιμέναμε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρο, οποιοδήποτε εταίρο, όποιου είδου συμφωνία και να είχαμε, ακόμα και συμφωνία EPA, ε, προστασία των επενδύσεων. Ξέρω ότι η χώρα σα στην ε, Ιταλία είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Το ρύζι είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν. Το ρύζι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο προϊόντων για του εξή λόγου και ξέρω ότι περιμένετε εδώ γιατί με ρωτήσατε. Βάσει του κανονισμού και γενικευμένων προτιμήσεων, ε, οι εγγυήσει για τι γενικευμένε προτεήσεις εξυπηρετούν συγκεκριμένου σκοπού ε, και ε, έχουν να κάνουν με επιτακτικέ ανάγκε ε, κατεπίγουσες για την οικονομική κατάσταση κάποιου μέλους που λαμβάνει την, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Αυτή είναι η νομική κατάσταση. Βλέπετε ότι είναι πολύ νομικίστικα όλα αυτά τα πράγματα, αλλά η διαδικασία προσωρινής απόσυρσης που ή αναστολή που εγκρίναμε για την Καμπότζη είναι ε, αυτό που του ζητάμε, η υποχρέωση να συμμορφωθούν. Πάντως δράση αναλάβαμε. Το κολέγιο των Επιτρόπων αναλάβει δράση για την ε, Καμπότζη και τους καλούμε να σκεφτούν τι θα γίνει με το ρύζι, αυτά που έχουν γίνει αρχικά. Θα δούμε μήπως το θέμα πάρει κάποια άλλη τροπή και επιληθεί. Για την Κίνα. Πρέπει να επιταχύνω, το βλέπω, μου το λέτε, Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε όμω να ολοκληρώσουμε την Κίνα, θα είναι πολύ δύσκολο να αποσπάσουμε συμφωνία με το τέλο του καλοκαιριού με την Κίνα. Διότι θα υπάρξουν ε, πολλέ καθυστερήσει ε, και όλο ένα κυρώνονται συναντήσει. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο η ταχύτητα. Θα πρέπει να είναι όριμε οι συνθήκε για να υπάρξει συμφωνία με την Κίνα. Και θα έχουμε την καταλληλότερη δυνατή συμφωνία. Πάντω με την Κίνα ε, επιτελείται κάποια πρόοδο. Και θα προχωρήσουμε όπως προχωρούμε και με τη ΣΥΠΑ. Έτσι έχουν τα πράγματα προς στιγμή. Το Brexit είναι ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τα πάντα. Είχαμε ε, μια συμφωνία με, στην πρώτη φάση και μια πολιτική δήλωση από κοινό με τον Μένο Βασίλειο, καλή την πίστη. Όταν ε, συνάπτηκαν μια συμφωνία, θέλει να την τιμήσει κιόλα, θέλει να τη σεβαστεί. Η συμφωνία αποχώρηση είναι ε, νομικώ έγκυρη και δεν υπάρχει τρόπος να πάμε προς τα πίσω, ε, ούτε εμείς, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλιώς θα πρέπει να παραβάσει διαδικασίες κατά του οποιοδήποτε πασπίστε το ανάποδο, ε, το αντίθετο. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και ποιους στόχους θέλουμε να πετύχουμε με τη μελλοντική συμφωνία. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Οι δηλώσει που έγιναν προσφάτω από διάφορου εκπροσώπου τύπου, υπουργού, πρωθυπουργού για του ίσους όρου ανταγωνισμού, είναι πολλέ και αντικρώμενε. ο κόσμο του Ηνωμένου Βασίλειου βιβλίο, είναι έντιμο και κρατάει το λόγο του. Ε, αν λοιπόν δεσμευτούν για κάτι, πιστεύω ότι θα το εφαρμόσουν. Ε, το έγγραφο μα ενδιαφέρει να δούμε ότι κάτι θέλουν. Σε πνεύμα λοιπόν για σκοπού καλή συνεργασία και καλή πίστη, ελπίζουμε ότι το Μένο Βασίλειο θα κοιτάξει να έχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόζει όσα υποσχεθεί. Τώρα, η εντολή του Συμβουλίου θα προκύψει, την, θα εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε πολύ αυστηροί εκεί ω προ του ε, όρου ανταγωνισμού, γιατί το ΕΒ είναι τεράστια αγορά και είναι και δίπλα μα. Ε, δεν είναι μακριά όπω Αυστραλία και ο Καναδά. Ξέρω ότι οι Καναδοί θα θέλαν πολύ να έρθουν κοντύτερα και αυτό ακούγεται πολύ στα βρετανικά μέσα, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που μα αρέσει. Ε, γιατί η συμφωνία με τον Καναδά θα μπορούσε να είναι ένα λιθαράκι για να πάμε σε μια καλύτερη συμφωνία ε, ή αυτό που θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντω, την επόμενη εβδομάδα θα προκύψει η εντολή, θα ολοκληρωθεί. Θέλουμε 2 Μαρτίου να ε, αρχίσουν οι διαπραγματεύσει και θα υπάρξουν 10 γύροι. Μέχρι το τέλο του Ιουνίου, ο κύριο Τζόνσον, ο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να αποφασίσει τι μετάβαση θέλει. Λέω δεν θέλει την περίοδο. Αν όμω τελικά τη θελήσει, ε, αν δεν τη θελήσει, θα πρέπει να έχουμε συμφωνία μέχρι το τέλο Οκτωβρίου. Ε, γιατί και το Κοινοβούλιο και άλλοι ε, άλλε πολιτικέ δομέ πρέπει να πούνε να συμφωνούν, διαφωνούν και ε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό παραθυράκι που μα υποχρεώνει να δώσουμε προτεραιότητα στα 10 κεφάλαια διαπραγματεύσεων με τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε. Αυτά είναι τα θέματα που έχουμε μπροστά μα και αυτά είναι τα διάφορα κεφάλαια. Τώρα, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, πάρει απόσταση από του κανόνε και τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο πιο πολύ αποκλίνει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι γραφειοκρατικός, ε, διοικητικό άχθος, ε, τη συμφωνίας. Πάντω, να κάνω την εξή παρατήρηση. Διότι νομίζω τα κράτη-μέλη καλό θα ήταν αυτό να το αντιμετωπίσουν κατάματα. Έχουμε ήδη μια συμφωνία. Πράγμα που σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετέχει από 31 Δεκεμβρίου 2020 ε, τα, στην εσωτερική αγορά και την Ελληνική Ένωση. Όμω ε, ε, έτσι κι αλλιώ θα αλλάξουν τα πράγματα από τον Γενάρη. Δεν ξέρω αν τα κρατημέλη κάνουν αρκετή προσπάθεια για να ενημερώσουν του συμμετέχοντε στην αγορά για το ποια θα είναι η αλλαγή στην καθημερινότητά του από 1η Ιανουαρίου 2021. Πρέπει στα κάτι μέλη να γίνει η ιανουαριου 2021 πρεπει στα κατι δουλειά και να του πούμε ότι η κατάσταση έχει ήδη αλλάξει, ακόμη και με αυτή τη συμφωνία. Ε, θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχαμε καμία συμφωνία, αλλά ακόμη και να υπάρξει συμφωνία που επιδιώκουμε, από άποψη επιμελητία διοργάνωση, από το πώ ε, διοργανώνουμε τι εμπορικέ μα σχέσει, πώ ταξιδεύουμε, θα υπάρξει τεράστια αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε ούτω ή άλλω καταλήλω. Για τον ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποβάλει, όπω είπα προηγουμένω, προτάσει, προτάσει προ εξέταση. 16 κάτι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί μα σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε καταρτήσει μια διαδικασία ώστε να έχουμε μια ε, ενδιάμεση και πολυμερή ομάδα συζήτηση, ένα πάνελ. κοιτάζουμε να γίνει και κάποια ε, μεταρρύθμιση αλλαγή στο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ και τις ερχόμενες εβδομάδες θα κοιτάξουμε αν μπορεί να υπάρξει ένα έγγραφο ουσίας με νοήματος για το δευτεροβάθμιο δικαιωτικό εργαλείο, ε, όργανο ως τον Ιούνιο τουλάχιστον. Ε, τα έχω θέσει αυτά και στις συζητήσεις μου με τις είπα. Δεν έχω πάρει απάντηση ακόμη, όμως μόλις πάρω θα σας πω ε, για την Ταϊβάν. Έχω πάρει... Έχω πάρει πληροφορίες από τον κύριο Χάντσεν. Έχω πάρει κάποιες πληροφορίες από τον κύριο Χάντσεν για την Ταϊβάν. Ναι, τη βρήκα, τη φυλάδα. Το μόνο που μπορώ να πω για την Ταϊβάν είναι ότι υπάρχει ε, διασύνδεση ανάμεσα στι διαπραγματεύσει που κάνουμε με την Κίνα και με την Ταϊβάν. Γιατί η λογική επενδύσεων στην Ταϊβάν είναι ότι θα έχουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα ανεφοδιασμού ε, μεταξύ Κίνα και Ταϊβάν. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα κομμάτι χωρί το άλλο. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα κάνουμε με την Κίνα ε, μέσα στο 2020 πριν προχωρήσουμε την Ταϊβάν αν προχωρήσουμε με την Κίνα, σίγουρα θα προχωρήσουμε και με την Ταϊβάν και αντίστροφα. Για την ε, συμφωνία που έκανε οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Κίνα, για την πρώτη φάση όπως λένε, η κυρία Χούμπνερ ρώτησε αυτό το πράγμα, έχουμε πει δημόσια ότι είναι ε, μία συμφωνία που δεν νομίζω ότι θα συμπορφούνται με τον ΠΟΕ, αλλά την αναλύουμε αυτή τη στιγμή ε, και αυτή είναι η αρχική μας άποψη. Θα φτάσουμε συμπεράσματα όμως ε, τις επόμενες εβδομάδες για να δούμε αν όντως ε, δεν συμμορφούνται με τον ΠΟΕ, αλλά έτσι μοιάζει εκ πρώτη όψεω, εκ πρώτη ανάγνωση. Ο κύριο Κέλλη ρώτησε για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και πλάς, αν θα συνεχιστεί μετά το 2023. Ε, το πιστεύω, γιατί γίνεται πολύ καλή δουλειά ε, με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και τέλη του επόμενου χρόνου θα αρχίσουμε τη διαδικασία για να δούμε αν το Κοινοβούλιο και μαζί με του συμφεροντούχου και του stakeholders, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το συνεχίσουμε. Ε, ελπίζουμε να ανανεωθεί έτσι όσο έχει, αλλά να βελτιωθεί το GSP+. Κλέρ ε, ρώτησε για το Μερκοσούρ. Ντέλι. Υπάρχουν θέματα για το πολιτικό κεφάλαιο που πρέπει να διευκρινιστούν με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και φυσικά αυτό θα πρέπει να σωματωθεί στη γλώσσα Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, είπαμε ότι απέναντι στους τομέες πολιτείες δεν ε, μειώνουμε τα πρότυπα. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε συμφωνία ε, με την Boeing και την Airbus με τους Αμερικανού. Ε, ορισμένοι λένε να περιμένουμε το, το αποτέλεσμα της, ε, του σώματο Προσφυγών τον Ιούνιο. Εγώ δεν συμφωνώ. Ε, σε αυτέ τι διαπραγματεύσει προσπαθούμε να βάλουμε κάποιε δεσμεύσει από του Αμερικανού για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ γρήγορη διαπραγμάτευση αν υπάρχει η πολιτική θέληση από του Αμερικανού γι' αυτό. Προσπαθούμε εμεί, από την πλευρά μας. Ε, το γεγονό ότι δεν αυξήθηκαν οι δασμοί πέρα από τα προϊόντα Airbus ε, την περασμένη Παρασκευή νομίζουμε ότι είναι καλό σημάδι ότι τη γλίτωσε ο γεωργικός τομέας και ο αμπελονικός τομέας. Έχουμε, πριν φύγω από το γεωργικό κομμάτι, έκανα αλλαγέ ούτω ώστε ο ίνος να στηριχθεί από τα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα. Αλλάξαμε κάποιου του κανόνε και τι συνθήκε, ούτω ώστε να έχει πρόσβαση ο ίνο ε, σε αυτή τη στήριξη. Η Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση θα σα δώσει περισσότερε πληροφορίε για τον αμπελοϊνικό τομέα. Αλλά τότε, όταν είχα κάνει αυτές τις αλλαγές, ο κλάδος τις υποδέχτηκε θετικά. Ε, δεν νομίζουμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην αγορά, αν ταραχεί στην αγορά. Ε, δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αν όμως υπάρξει αναγεραρχή στην αγορά, ε, θα τα έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μα. Ίσως η Γαλλία όμω, ή οποιαδήποτε άλλη πληττόμενη χώρα θα μπορούσαν να ζητήσουν ε, τη χαλάρωση των ε, κρατικών ενισχύσεων για να στηριχθεί ο εινικός τομέα και οι επιχειρήσει αυτέ. Χωρί να χρειάζεται να περάσουμε από τι δομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πιστεύω ότι αυτή η ιστορία που έχει γίνει με την Κίνα ε, θα διατηρηθεί παρά τις προσπάθειες των Αμερικανών ε, σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις. Η Κινέζη μας είπε ότι η συμφωνία του Νοεμβρίου ισχύει. Perfect, uh, Τέλεια, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, εκτεταμένη απάντηση των 20 ερωτήσεων και των σχολείων. Νομίζω ότι πλέον έχουμε μια σαφή εικόνα για την ε, ε, μελλοντική εμπορική πολιτική της Ένωσης και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα είμαστε σε επαφή ε, για το θέμα της κοινής μας δουλειάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. So, Όποιος αποχωρήσει, παρακαλώ να αποχωρήσει ήσυχα. Περνάμε στο θέμα 13 της ομάδας παρακολούθησης. Πρώτα θα έχουμε την αναφορά της ομάδας της Ελβετίας. Yes, thank you. the monitoring group for the... Ευχαριστώ. Οι ομάδες παρακολούθησης των χωρών ΕΖΕΣ δεν είναι μόνο η Ελβετία, είναι και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενστάιν. Έγινε δεύτερη συνάντηση στις 22 Ιανουαρίου Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον Γενικό Γραμματέα της ΕΖΕΣ, τον κύριο Γκετάς, όπως επίσης ε, τους αναπληρωτές Εγεχόφ και Λούθερσον. Έκαναν μια παρουσίαση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω της Συμφωνίας ε, ΕΖΕΣ εοχό, τις ε, ευθύνες της, της γραμματείας ΕΖΕΣ και μια επισκόπηση του δικτύου ελεύθερου εμπορίου. Φέτος η ΕΖΕΣ ε, ε, ε, ε, γιορτάζει την 60η της επέτειο, ενώ η ΟΕΟΧ γίνεται 25. Ε, ε, επίσης η Βρετανία φεύγει και από τον ΕΟΧ. Ε, τα κράτη ΕΖΕΣ ΕΟΧ προετοιμάζουν τη δική τους συμφωνία ε, ε, αποχώρησης αλλά προετοιμάζονται και για μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία. Επίσης συζητήθηκαν οι μελλοντικέ σχέσεις με την Ελβετία, το θέμα της ελεύθερης διακίνησης των ατόμων και τη συμμετοχή στην αγορά. Ε, το, έγινε το Μάιο δημοψήφισμα για το θέμα της ελεύθερης διακίνησης και δεν θα υπογράψει τη συμφωνία πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελβετία μέχρι ότου α, θα γίνει το ε, δημοψήφισμα, συγχωρείτε, και μέχρι τότε δεν θα υπογραφεί. Είναι επίση σαφέ ότι οι συζητήσει για το Mercosur είναι θέμα που αφορά και τι χώρε ΕΖΕΣ. Έχουν και αυτέ καταλήξει σε συμφωνία που πρέπει τώρα να κυρωθεί και βεβαίως υπάρχει συζήτηση στις τέσσερις αυτές χώρες, κυρίως Νορβηγία και Ελβετία και λιγότερο Λιχτενστάιν και Ισλανδία. Επίσης συζητήσαμε για την κατάσταση στον ΠΟΕ και πώς οι χώρες ΕΖΕΣ επέλεξαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή με τρόπο διαφορετικό σχετικά με την ε, ενδιάμεση συμφωνία επίλυσης ε, ε, προσφυγών και τώρα ε, ε, ε, από την, από την συνάντησή μας, εκτός από την Ορβηγία, εντάχθηκε και η Ελβετία σε αυτή τη συμφωνία. Επίσης, δύο λόγια για τις μερίς συνομιλίες Ελβετίας, είπα, για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, η οποία δεν προχώρησε πολύ μέχρι τούδε. Η επόμενη ομάδα επιτήρησης θα συνεδριάσει στις 18 Μαρτίου, οπότε φυσικά θα σας προσκαλέσουμε, θα στείλουμε και την η ε, ημερήσια διάταξη και ελπίζω να συναντήσω τους ε, νέους σκιώδες ε, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Όχι. Οπότε περνάμε στην επόμενη. Είπατε, αναφερθήκατε στο Μερκοσούρ, κύριε Βόμπορν, και η επόμενη είναι η Μερκοσούρ, Ο κύριος Κάνας θα μας κάνει μια παρουσίαση. Ευχαριστώ. Μου λένε ότι μιλάω πολύ γρήγορα, ότι είμαι πύραυλος <laughs> για την ομάδα παρακολούθησης του Μερκοσούρ. Πάντα μου το λένε, Πρέπει να μειώσω λίγο ρυθμούς, να κατεβάσω ρυθμούς. 22 Ιανουαρίου κάναμε την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης Μερκοσούρ, που μας επέτρεψε να κάνουμε μία πρώτη προσέγγιση, approach, για την κατάσταση της συμφωνίας. Ε, η συγητής ήταν η Σάντρα Γκαλίνα, βασική διαπραγματεύτρια για τα εμπορικά και η κυρία Λορένθο για τα πολιτικά στοιχεία του Μερκοσούρ. Έχουμε υπογράψει το εμπορικό κομμάτι 20 Ιουνίου του 2020. Τώρα για το πολιτικό κομμάτι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα. Για την ολοκλήρωση του εγγράφου, είμαστε στην νομική αναθεώρηση της συμφωνίας από ό,τι μας λένε οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Έχουμε ενδείξεις για το πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν το κείμενο για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. μπορούν να περάσουν, λέει, έξι μήνες με ένα χρόνο. Μπορεί και περισσότερο. Μας είπαν ότι, ε, μία φορά μας λένε έξι μήνες, μετά μας λένε οχτώ μήνες, μετά μας λένε ένα χρόνο. Κάτι τέτοιο. Αυτό μας είπε. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι μπορούμε να το κλείσουμε. Έχουμε μία ακρόαση στην Επιτροπή Ίντα, 29 και 30 Απριλίου. Θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε το πάνελ, ούτως ώστε να είναι όσο πιο ενδιαφέρουσα η ακρόαση, στην ακρόαση θα πρέπει να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις πάνω στη συμφωνία, θετικές, αρνητικές για το εμπορικό κομμάτι της συμφωνίας. Θέλουμε να είναι πλούσια η συζήτηση, να επιτρέψει μια πραγματικά σοβαρή, ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση για τη συμφωνία αυτή. Επίσης, η Επιτροπή θα στείλει ε, στο Μερκοσούρ, θα πάει, θα ταξιδέψει στο Μερκοσούρ την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Το Monitoring Group θα συνεδριάζει περιοδικά. Θα έχουμε συνεδριάσεις για να συζητάμε συγκεκριμένα θέματα ή συγκεκριμένα κεφάλαια. Θα διαιρούμε, ας πούμε, σε θεματικές ενότητες το τη συμφωνία και θα κάνουμε συζητήσει, ούτω ώστε να έχουμε τι περισσότερε δυνατέ πληροφορίε πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Και θα γίνει αυτή η συζήτηση πριν γίνει η τελική συζήτηση. Αυτά, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομάδα παρακολούθησης, Μαρόκο. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση στις 22 Ιανουαρίου. Ήταν, ε, ήταν ε, μάλιστα σχετικό με την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε εδώ στην Επιτροπή και είχαμε και συζήτηση για τη συμφωνία με τη Δυτική Σαχάρα και τα σχετικά προϊόντα. Ήταν η πρώτη συνάντηση αυτή τη ομάδα παρακολούθηση και προσκληθεί και η ΕΕ για να κάνει κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει για τι πολιτικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου και επειδή η καθήλυνα αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Ταξούντ, είχαμε μια διεξοδική παρουσίαση για το μηχανισμό. Το μηχανισμό που επιτρέπουν στις τελωνιακές αρχές να έχουν πρόσβαση ε, και τα προϊόντα που έρχονται από τη Δυτική Σαχάρα. Ε, τα στοιχεία ήρθαν ε, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουν και θα πρέπει να έρχονται και σε μηνιαία βάση. Η Γενική Διεύθυνση προβλέπει ότι το Μαρόκο ε, δίνει αρκετέ ε, πληροφορίε με του συστήματο που δεν έχουν δώσει ω τώρα άλλοι εμπορικοί εταίροι. Το δεύτερο θέμα ήταν η κατάσταση εμπορικών διαπραγματεύσεων με το Μαρόκο και είναι γεγονό ότι το Μαρόκο ανέστηλε τι εμπορικέ διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Η Γενική Διεύθυνση Trade μας ενημέρωσε για τις πρόσφατες συναντήσεις με μαροκινούς υπουργού ε, εμπορίου και πώς μπορεί να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει. Το Μαρόκο θα ήθελε να κάνει μια σειρά από μελέτες αντικτύπου και να εξυγχρονίσει τις ε, συμφωνίες βάσει της νέας εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τρίτο θέμα που συζητήσαμε ήταν η κατάσταση του πώς έχουν τώρα γεωγραφικές ενδείξεις στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Το παρόν κείμενο έχει κολλήσει στο Συμβούλιο γιατί δεν μπορούν να εντοπίσουν την εδαφική ε, ισχύ της συμφωνίας κάτι που για την ώρα δεν καλύπτει το έδαφος της δυτική Σαχάρας. Um, Ευχαριστούμε. Για το Μεξικό, Ήμα. Στο Πρόεδρε, θέλω να ενημερώσω όλους ότι ξέρουμε ότι η συμφωνία με το Μεξικό είναι μια συμφωνία εξυγχρονισμού. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκαν. Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 περιμέναμε, ούτως ώστε να έχουμε μια προσφορά ε, από το Μεξικό για τις ε, προσφορές που μας κάνουν σε πολιτιακό επίπεδο για τις υπεργολαβίες. Τον Ιούλιο του 2018 έγιναν εκλογές στο Μεξικό. Εν συνεχεία, το 19 έγιναν εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, την τελευταία δέσμευση που έπρεπε να αναλάβει το Μεξικό ε, για, την, για το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων ε, των, σε πολιτιακό επίπεδο έπρεπε να το ανοίξει στις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πρέπει να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις του και τις προϋποθέσεις τόσο ώστε να, παρουσιάσαμε, να παρουσιάσουμε τη συμφωνία προς σύμφωνη γνώμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια συμφωνία, επαναλαμβάνω, εξυγχρονισμού, που πάει πολύ πιο πέρα από την αρχική συμφωνία ε, που υπογράφηκε το 2000, που συνήθι το 2000, που ήταν η πιο ε, φιλόδοξη συμφωνία τότε. Και ελπίζουμε και η σημερινή συμφωνία να είναι, να είναι φιλόδοξη για την αγορά μας και για την προσπάθεια που κάνει το Μεξικό για να προβεί σε βιώσιμη ανάπτυξη, για να σεβαστεί τα εργασιακά δικαιώματα. Έπρεπε να υπογράψει μια, μια πολύ σημαντική σύμβαση, την υπαριθμό 98 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το έκανε. Έχει επίσης 340 γεωγραφικές ενδείξεις που δεν ανήκουν ε, σε αυτό το πλαίσιο με το οποίο δουλεύουμε για τα γεωργικά προϊόντα. Πρέπει επίσης ε, να σεβαστεί το δημόσιο σύστημα προστασίας των επενδύσεων. Ένα από τα στοιχεία που τόνισε το Monitoring Group και που μας είπε η, ο κύριος Ματίας Γιόρενσε, που είναι υπεύθυνο για την Εθνική Αμερική, μίλησε για την διαφάνεια και τις πληροφορίες που έχει στην ιστοσελίδα της Οικομισιόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πρόκειται για μια συμφωνία πολιτικής σύνδεσης και δεν έχουν πληροφορίες για το κομμάτι που αφορά τα θέματα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, για την ΑΦΕΤ και για, την, για τα όσα ενδιαφέρουν τη ΛΥΜΠΕ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξανατονίζω τη σημασία που έχει διαφάνεια. Ε, η διαφάνεια δεν είναι μόνο τμήμα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφορά όλα τα θέματα. Όταν μιλάμε για μια ε, πολιτική εμπορική συμφωνία, και μάλιστα εδώ πέρα έχουμε και μια πολιτική συμφωνία συνεργασίας, είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια σε όλη την συμφωνία. Ερωτήσεις. Κάθλιν, ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν είμαι συγγήτρια, όμως η συγγήτρια ήταν η Νικολά Τάντε που δυστυχώς μας έφυγε, αλλά ελπίζουμε να επιστρέψει στη διπλανή ομάδα. Με μεγάλη χαρά όμως θα σας ενημερώσω λίγο για την ε, ομάδα παρακολούθησης. Στις 18 ε, Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη ε, συνάντηση, η 28 Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη συνάντηση στις Βρυξέλλες. Ε, είχαμε δύο μέρη. Πρώτα μια ενημέρωση με τον κύριο Κάινερ, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ένωσης και μετά υπήρχε ένας ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών για να παρουσιάσει τις δικές τους προτεραιότητες της διαπραγματεύσης Η ενημερώθηκε εκτεταμένα η ομάδα για τις ε, διαπραγματεύσεις για τον Νοέμβριο, τη συνάντηση στο Νταβός και τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων εν ώψη της Υπουργικής του ΠΟΕ ε, στον Ουσουλτάν. Οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις είναι επικοδομητικές με την ενεργό συμμετοχή πολλών κρατών, τώρα 83, μεταξύ των οποίων πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι ε, πολύ ενθαρρυντικό ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί εταίροι σε αυτή τη, στην σημαντική πολυμερή ε, εμπορική πρωτοβουλία. Και επίσης πολλές άλλες, ε, πολλοί άλλοι γύροι διαπραγματεύσεων σχεδιάζονται που είναι σημαντικές, σημαντικοί για να μπορέσει να επέλθει ουσιαστική πρόοδο σε, κάποια από τα θέματα που καλύπτει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Επίτροπος, κάποια πρόοδο σημειώνεται, αλλά δεν έχει, θα υπάρξει συμφωνία για τον ενόψη του Νουρ Σουλτάν. Ερωτήσεις όχι, οπότε ε, ανατολικές ε, ε, ε, ε Εταιρική σχέση Ανατολικής και Νότιας Αφρικής. Στις 28 Ιανουαρίου έγινε μια ενημέρωση από την κυρία Σεσίλ Μπιγιό, επικεφαλής ε, του Τμήματος ε, Οικονομικών Εταιρικών Σχέσεων για την Αφρική, Καραϊβική και τον Ειρηνικό και τι ε, υπερπόντιε χώρες και εδάφη μετά έγινε ο δεύτερος γύρος στις 15 και 17 Ιανουαρίου στις Σεϊχέλες και η πρόοδος ε, ε, και συζητήθηκε η πρόοδος για την, ε, για την εκτίμηση των επιπτώσεων των, της βιωσιμότητας. Μετά έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, στις 28 Ιανουαρίου έγινε η συνάντηση σε σχετικά με το ταξίδι του κυρίου Χόγκαν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, η επιθυμία ήταν να αποκλιματοκωθεί η κατάσταση και να γίνει μια προσπάθεια εξέβρεσης ε, κάποιας συνεννόησης για κάποια θέματα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Όσον αφορά τη Χιλή, υπήρξε μια επιτροπή παρακολούθησης ε, η κυρία ε, Ραφαέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έγινε η πρώτη ομάδα ε, συνεδρίαση στις 29 Ιανουαρίου φέτος με ενημέρωση από την κυρία Εύα Μαρία Καρμπατιέρα, ε, αναπληρώτρια επικεφαλής της Μονάδας Λατινικής Αμερικής της Γενικής Διεύθυνσης Trade, η οποία μας έδωσε, μας την κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον εξυγχρονισμό του πυλώνα του εμπορίου, της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής ενημερωτικά δεν, δεν λειτουργεί ε, ε, όπως αναμενόταν λόγω των νέων παγκόσμιων προκλήσεων και μετά από έξι γύρους διαπραγματεύσεων πλέον ε, θα επιτευχθεί ή ακόμα πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, γεωγραφικών ενδείξεων, το, θέματα επενδύσεων ενέργειας και πρώτων υλών και το εμπόριο του εμπορίου ε, ήταν μια θετική αξιολόγηση. Προχώρησε παρά ε, την κατάσταση στη Χιλή. Είμαι αισιόδοξη και θεωρώ ότι εν γέννη αυτή ήταν η εντύπωση, ότι δηλαδή το νέο αυτό κοινοβούλιο μπορεί να ε, γνωρίσει την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Να το ευχηθούμε. Επίσης ε, προσπαθούμε να πετύχουμε ε, το βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χιλή μέσω μια ε, εξυγχρονισμένης τέτοια συμφωνίας, θέματα δικαιώματα των αυτοχθόνων, θέματα φύλου και επίσης τη υπογράμμισα την ανάγκη να υπάρξουν, ε, υπάρχει συμβελτίωση θεμελιωδών δικαιωμάτων των αυτοχθόνων στην ε, Χιλή. Στις 26 Απριλίου θα υπάρξει κάτι μια, κάτι ως ανταπόκριση της, ε, των διαμαρτυριών του 2019. Ο επόμενος γύρος θα γίνει τον Απρίλιο-Μάιο, κάτι τέτοιο. Ε, Άρα θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ ενδιαφέρον διάστημα για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εφόσον δεν έχουμε κάτι παραπάνω, η Ιαπωνία. Άμεσα, χωρίτε. Είμαι πρόεδρος της ε, διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με τη Χιλή. Είχε προβλεφθεί η χιλή στην μπλε εβδομάδα του Οκτώβρη, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε στη χιλή. Για λόγους ασφάλειας δεν μπορέσαμε να πάμε στη χιλή, προφανώς. Το Φεβρουάριο δεν μπορούμε να πάμε στην Τυρκουάζ εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην Χιλή τον, το μήνα αυτό είναι τα πάντα κλειστά. Είναι σαν Αύγουστο εμάς και θα πάμε τελικά 4 με 6 Μαρτίου. Θα έχουμε μία αποστολή 9 ευρωβουλευτών από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς είναι η κατάσταση στη Χιλή, γιατί επιπλέον στις 26 Φεβρουαρίου ξεκινάει η προεκλογική εκστρατεία εν ώψη του δημοσκοπίσματος που θα γίνει στις 26 Απριλίου. Ε, είναι σημαντικό να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν. Πολύ συναρπαστικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε κύριε Λατσίνη για την Ιαπωνία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η ομάδα παρακολούθησης ΣΥΝΤΑ για την Ιαπωνία μας επέτρεψε να έχουμε μια πρώτη θετική αποτίμηση της εφαρμογής της ε, Συμφωνίας ε, Εταιρικής Σχέσης, Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με την ε, Ιαπωνία κοιτάξαμε τις πρώτες πτυχές εφαρμογής της συμφωνίας από την 1η Φεβρουαρίου του 2019 και είδαμε και κάποια αριθμητικά στοιχεία σε ποσοστά διψήφια. Είδαμε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τις εμπορικές ροές ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στο διεθνές προσκήνιο. Ε, υπογραμμίστηκε ότι τα ωφέλη της συμφωνίας αυτής ξεπερνούν την άρση των διασμολογικών φραγμών για τα προϊόντα. η ε, μη δεσμολογική φραγμή, το άνοιγμα των αγορών για τις δημόσιες προμήθειες ε, των δημόσιων υπηρεσιών είναι σημαντικά αποτελέσματα που φέρνουν ωφέλη για τις οικονομίες και των δύο περιοχών. Ήταν θετική στάση των Ιαπωνικών αρχών, γιατί κάθε φορά που χρειάζεται να ασχοληθεί με τα θέματα της υλοποίησης, τη εφαρμογή των κανόνων, το αντιμετωπίζουν θετικά. Ειδικά η Γενική Διεύθυνση Ταξούν ανέφερε τις ε, τελωνιακέ ε, διαδικασίες σε σχέση με τις γραφικέ ενδείξει και την αντιμετώπιση των ε, ε, δασμολογικών ε, διαφορών για να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ενημέρωσε ότι προβλέπεται συνάντηση του Επιτρόπου Χόγκαν με τον Υπουργό, με τον Ιάπωνα Υπουργό Εμπορίου, για να δούμε το πολιτικό πλαίσιο. Κατά τη συζήτηση είδαμε μια-δυο συγκεκριμένε ερωτήσει για τον αντίκτυπο τη μικρομεσαία επιχειρήση την κατάσταση προόδου των βασικών ε, συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την εργασία και την απασχόληση και την προστασία των επενδύσεων, ιδίω για, για την παραγωγή τροφίμων που είναι πολύ ε, ενδιαφέροντα και σημαντικά στο πλαίσιο του πυρηνικού ατυχήματος της Φουκουσίμα. Η ομάδα παρακολούθησης ΙΝΤΑ για την Ιαπωνία θα συνεχίσει να παρακολουθεί ε, την ε, υλοποίηση της συμφωνίας και θα δούμε τα στοιχεία που μπορεί να χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία ακούγεται όλο αυτό. Ερωτήσεις. Κύριε Βίνκλερ, για την Κίνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Στις 5 Φεβρουαρίου είχαμε την ομάδα παρακολούθησης, ε, ε, τη συνάντηση της ομάδας παρακολούθησης για την Κίνα επικεντρωθήκαμε σε δύο διαφορετικά θέματα. Πρώτα απ' όλα, επισκόπηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και θεματολόγιο το 2020. Την, ε, τον κατάλογο προτεραιοτήτων μας δηλαδή. Επ' αυτού έχουμε σημαντικού, σημαντικές συνόδους κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας πρώτα απ' όλα στα τέλη Μαρτίου την ε, σύνοδο για να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό και τα σχετικά μέτρα που μπορεί να έχουν αναλυθεί. Και μετά το Σεπτέμβριο έχουμε και την ειδική σύνοδο που θα την υποδεχτεί η Γερμανία ως προεδρεύουσα στο Συμβούλιο τότε και θα έχουμε πολλές ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις εντατικές ε, πλαίσιο συνεργασίας, περιβαλλοντικές ενιστώσεις και σχετική συνεργασία. Οι δύο σύνοδοι, λοιπόν θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να παρακολουθήσουμε στενότερα τα θέματα αυτά. Όπως είδαμε στο διάλογο με τον Επιτρόπο Χόγκαν νωρίτερα σήμερα, στην ομάδα παρακολούθησης και σε εμά δηλαδή, ασχοληθήκαμε πολύ και με τη Συμφωνία Γεωγραφικών Ενδείξεων, την οποία συνήψαμε πρόσφατα με την Κίνα και τη φάση υλοποίηση της συμφωνίας αυτής. Επίσης, το θέμα του ενδεχόμενου αντικτύπου Ή το τι θα γίνει με την ε, ενδεχόμενη συμφωνία ΙΠΑ ε, Κίνα φάση 1 ή την συμφωνία γεωγραφικών ενδείξεων με την Ιαπωνία. Αναπτύχθηκαν πολλά ενδιαφέροντα, τα ακούσαμε και τον Απίτροπο Χόγκαν. Η Γενική Διεύθυνση Agri και Trade είναι αρκετά ε, Πιστεύουν ότι η συμφωνία με τι γεωγραφικέ ενδείξει έχει τις κατάλληλε διατάξεις για να υπερισχύσει σε σχέση με αυτό το είπαμε την Κίνα. Δεύτερο θέμα ήταν το πώ προχωρούν οι διαπραγματεύσει ε, για την ε, σφαιρική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα για τις επενδύσεις. Εκεί υπήρχαν ε, νέα και καλά και κακά. Δύο γύρω έχουν οργανωθεί. Επιτροπή αξιολογεί θετικά την ε, προθυμία των Κινέζων συναδέλφων να συνεργαστούμε. Όμω η προσφορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Κίνα είναι πολύ φιλοδοξότερη από την αντίστροφη, την προσφορά των Κινέζων προ εμά. Χρειάζεται περισσότερη ελαστικότητα για τι ε, επενδύσει και βεβαίω υπάρχουν ακόμα εκκρεμή ζητήματα. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, η ε, διαφάνεια, οι βιομηχανικέ επιδοτήσει, η ε, βιώσιμη ανάπτυξη, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Η κατάσταση μάλλον δεν θα βελτιωθεί άμεσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί και τα επιδημιολογικά. Θα δούμε τι θα γίνει το Μάρτιο ε, στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας που μπορεί να οργανωθεί και με βίντεο ε, και τηλεδιάσκεψη. Ε, τέλος, και επειδή εγώ δεν μπόρεσα να προεδρεύσω στη συνάντηση, είχαν εγκλημένες υποχρεώσει. η κυρία ε, Ροντρίγκες Μιγγέλη είχε αναλάβει. Ε, αυτά μπορούσα να σας πω ως εδώ από πλευράς μου. Ευχαριστούμε. Ε, περνάμε λοιπόν στην τελευταία επιτροπή, Ουκρανία. κύριο Γιώρη, ευχαριστώ. Ε, γιορτάσαμε χτες ε, την ε, επέτειο της ε, Επιτροπής Παρακολούθησης χθες. Ενημερωθήκαμε Μιλάμε για την υλοποίηση της πρώτης ε, συμφωνίας σύνδεσης νέας γενιάς με τους εμπορικούς εταίρους που εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του 2014 από την Επιτροπή. Αυτή η EFTA ε, εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2016. Η Κομισιόν χαιρέτησε τη νέα κυβέρνηση του κ. Χελέντσκι και πιστεύει ότι η συνεργασία είναι ευκολότερη και πιο δυναμική. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ονόμασε τη νέα κυβέρνηση ένα καθεστώς τούρμπο και μοιάζει ότι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν τις ε, προηγούμενες, ε, τους προηγούμενους συμβιβασμούς, τις προηγούμενες συμφωνίες. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν σαφώς την θετική τάση. Οι εμπορικές ροές ποτέ δεν ήταν στα επίπεδα του 2019 προηγουμένως. Οι εξαγωγές της Ένωσης έφτασαν ε, επίπεδα ρεκόρ 28,8 εκατομμύρια ευρώ, ε, δισεκατομμύρια ευρώ ε, σε σχέση με το, είχαμε μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2014, αλλά και οι εισαγωγές έφτασαν ρεκόρ 19,8 δις ευρώ αύξηση κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άρα η συμφωνία αυτή αποδίδει, η διαδικασία βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί, πολλά πρέπει να γίνουν σε σχέση με την υλοποίηση, την εφαρμογή της και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της προσαρμογής λόγω των παραρτημάτων και η Ουκρανική πλευρά πρέπει να προσαρμοστεί στους εξελισσόμενους κανόνες μας. Η Κομισιόν ανέφερε τους βασικούς τομείς όπου έχει γίνει ε, πρόοδος, ε, δημόσιες ε, προμήθειες, SPS και τα τελωνία. Επεσήμανε κάποια κρεμή ζητήματα επίσης η Επιτροπή όπως η απαγόρευση εξαγωγών από την Ουκρανία, για το πάνελ εμπειρογνωμόνων και επίσης ε, καταφέραμε να λύσουμε διάφορα θέματα γρήγορα και να ε, ε, προχωρήσουν κάποια θέματα της νέας αυτής συμφωνίας. Η Ουκρανία μοιάζει ότι σκοπεύει να διευρύνει την επερχόμενη αναθεώρηση εμείς θα θέλαμε να παραμείνουμε στο υφιστάμενο πλαίσιο και θα δούμε. Αυτά ουσιαστικά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Αν όχι, προχωράμε. Κλείνοντας το σημείο 13, περνάμε στο 14 η προσωρινή απόσυρση του καθεστώσος, του καθεστώτος όλα εκτός από όπλα με την Καμπότζη. Έχουμε διαρθρωμένη συζήτηση με την Επιτροπή Όγκεν. Υπάρχει κατεξουσιοδότηση πράξη και τώρα έχουμε μια σύντομη παρουσίαση. Peter Burns. και ο κύριος Χάινου Μάριος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο πρέσβης της Καμπότζης, ο κύριος Νομ Πίσετ. Ε, καλώς ορίσατε. Πίτερ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Χόγκαν μίλησε ήδη. Να επεκταθώ λιγάκι. Η Καμπότζη, ε, με την Καμπότζη έχουμε την Οικονομική Συμφωνία εταιρική Σχέσης ε, και την απόσυρση από αυτήν. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών και να προωθήσουμε τα διεθνή πρότυπα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Ο σεβασμό των, δικαιωμάτων αυτών είναι ως λήθο των ε, ενωσιακών πολιτικών και μονομερείς ε, προτιμησιακές ε, συμφωνίες ε, όλα πλην των όπλων εφαρμόζονται υπό αυτές τις προϋποθέσεις. μετά από ένα χρόνο που έχουμε έρθει σε επαφή με τις αρχές της Καμπότζης, τελικά υιοθετήσαμε τον κανονισμό προσωρινά και Προς, ε, εν μέρη έχουμε αποσύρει τι ε, προτιμήσει για την Καμπόζη. Αυτή ο κανονισμό έχει διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ένα ε, επεξηγηματικό σημείωμα. Αυτή η απόφαση απόσυρση ε, δικαιολογείται γιατί έχουμε συστηματικέ και σοβαρέ ε, παραβιάσεις της κυβέρνησης Καμπότζη, των αρχών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχουν στο ε, σύμφωνο δικαιωμάτων και δεν υπάρχει πρόοδος στον τομέα αυτών από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία το Φεβρουάριο του 2019. Όταν λάβουμε την απόφαση για τη μερική απόσυρση των προτιμήσεων, η Κομισιόν ήθελε να διατηρήσει του στόχου ανάπτυξη του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε και τη μη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διατήρηση των στόχων ε, του εργαλείου GSP ω αναπτυξιακό εργαλείο, ε, δεν είναι καθόλου εύκολη προσπάθεια. Ε, η απόσυρση των α, προτιμησιακών δασμών ε, και η αντικατάστασή τους με τους κλασικούς δασμούς MFN θα επηρεάσει διάφορα προϊόντα, ζάχαρη κτλ. Έχουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ ε, που επηρεάζονται, ε, αξίας, εξαγωγές που επηρεάζονται από αυτό το σύστημα. Ε, εμείς θέλουμε με αυτό το σύστημά μας να υποστηρίξουμε βάρο της αναπτυσσόμενων χωρών για να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους ε, και να ενισχύσουν την παρουσία τους ε, στις διεθνείς αλυσίδε αξιών. Η Κομισιόν αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίζουμε ακόμα την οικονομική ανάπτυξη της Καμπότζης και την διαφοροποίηση των εξαγωγών τη. 80% των εξαγωγών συμπεριλαμβάνουν και τις αναδυόμενες επιχειρήσεις ε, βιομηχανίες, κάποια ε, είδη ρουχισμού και τρόφιμα θα, έχουν, ε, θα εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά ε, αδασμολόγητα. Ε, σκεφτήκαμε να αποσύρουμε τελώ τι προτιμήσει GSP και GSP+, όπως το κάναμε με τη Μιαμάρ, Σιλάνκα και Λευκορωσία. Αλλά η μερική απόσυρση θεωρεί η Κομισιόν ότι εξυπηρετεί το διπλό μα στόχο. Να υποστηρίξουμε τον λαό τη Καμπότζη και, και τη χώρα γενικά και να συνεχίσουμε το διάλογο με την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα παραβίαση των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων. Η BA, όλα πλην όπλα, ήταν σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των εξαγών τη Καμπότζη. Και αυτό συνέβη για την Καμπότζη τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση Καμπότζη είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 και πλασιάστηκαν ε, σε σχέση με το τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε τον κανονισμό εξιοδότηση μετά το, την θέτηση από το Σώμα των Επιτρόπων το Φεβρουάριο και θα πρέπει να πει την άποψή του. Το Κοινοβούλιο έχει τέσσερι μήνε για να αντιδράσει στον εξιωτικό αυτοκονισμό. Εάν δεν είσαστε αντίθετοι με το καθεστώς, τότε θα στις 12 Αυγούστου του 2020 θα τεθούν σε ισχύ τα νέα μέτρα. Παρά την απόφαση απόσυρση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ε, έχει σχέσεις με την Καμπότζη και να παρακολουθεί εκ του στην κατάσταση και για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και τα στεγαστικά δικαιώματα. Η πρώτη δημόσια αντίδραση της Καμπότζης είναι ότι η Καμπότζη, παραθέτω, είναι δεσμευμένη στην ενίσχυση περαιτέρω των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αμοιβαίου συμβασμού, ε, αμοιβαίων συμφερόντων και σεβασμού. Θα έχουμε την Κοινή Επιτροπή, είναι η επόμενη συνεδρίαση, που θα γίνει μέσα Μαρτίου του 2020 και η τελική ευθύνη για επανάκτηση των προτιμησιακών, ε, της προτιμησιακής πρόσβασης ε, στην ε, ενωσιακή αγορά με EBA, όλα πληνόπλα, είναι θέμα της Καμπότζης. Ελπίζουμε να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις η πλευρά της Καμπότζης και με τα ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα, τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάριος. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνεχίζει να έχει σοβαρές ανησυχίες για τα πολιτικά δικαιώματα στην Καμπότση. Τα τελευταία τρία χρόνια διαπιστώσαμε επιδείνωση του σεβασμού προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένου και του περιορισμένου χώρου της πολιτικής ε, αντιπολίτευσης των μέσων και των μέσων ενημέρωσης. Όπως προβλέπει ο κατεξουδότης διαγωνισμός για το θέμα των ε, εμπορικών προτιμήσεων, η Καμπότζη έχει κάνει σημαντικές δράσεις κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης του CNRP, του, ε, του Κόμματος Εθνικής Διάσωσης της ε, Καμπότζης, έχει περιερώσει τα εκλογικά δικαιώματα στη χώρα. Οι δράσεις αυτές συμπεριλάμβαναν συγκεκριμένα την σύλληψη του Κεμ Σόκα, προέδρου του CNRP, όπως επίσης και την διάλυση του CNRP και τις τροποποιήσεις ε, του κώδικα πολιτικών κομμάτων. Επ' αυτών, ελάχιστα έχουν αλλάξει από την, από την έναρξη της διαδικασίας ε, της απόσυρσης της ε, της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών τον Φεβρουάριο του 19 εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη η λειτουργία του CNRP και τα μέλη του συνεχίζουν να είναι ε, ε, ε, να διώκονται. Μετά την, δικαστική διάλυση, την διάλυση από τα δικαστήρια του βασικού κόμματος αντιπολίτευσης, η Καμπότζη έχει γίνει ένα μονοκομματικό κράτος και οι σχεδόν όλοι οι θέσεις ε, των εκλεγμένων μελών του CNRP μεταφέρθηκαν στο ε, κυβερνών κόμμα. Ο Κέμ Σόκχα ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου ε, συνελήφθη, ε, απελευθερώθηκε από τον κατοίκον περιορισμό αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν έχει απαλλαγή και δεν μπορεί να ασχοληθεί με οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα. Ο Ζώσεφ Πορέλ, ο υπατός εκπρόσωπος, συναντήθηκε με τον κύριο Κον τον Δεκέμβρη του 2019 στο πλαίσιο των, της συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών χωρών ΑΣΕΜ και ε, στο, με την ευκαιρία αυτή ε, έθεσε το θέμα του ότι η Καμπότζη πρέπει να ανοίξει το ταχύτερο δυνατόν το πολιτικό χώρο. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τους ερχόμενους μήνες θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την κυβέρνηση Καμπότζης και θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να ξεκινήσει η Καμπότζη μια δημοκρατική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης μέσω ε, ενός ειλικρινούς διαλόγου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο θα έχει ο εισηγητής και οι ισχυώδεις εισηγητές. Um, uh, Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ. Τα βλέπουμε και στην ομάδα παρακολούθησης ε, των σχέσεων με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Και βλέπουμε τη στάση έχει τηρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι η όλη συλλογιστική, είναι πολύ, το όλο σκεπτικό είναι πολύ ε, βάσιμο και πολύ καλό και το αποτέλεσμα, διότι ο σκοπός που επιδιώκει η Επιτροπή είναι σωστός. Η επιλεκτική και προσωρινή αναστολή είναι η σωστή κίνηση. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε την καταξιόδοξη πράξη, όμως ελπίζοντας ότι η Καμποτζιανή κυβέρνηση μπορεί να σκεφτεί ότι η ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει αυτή η κατεξοδότηση πράξη είναι 12 Αυγούστου ε, του 2020, μπορεί μέσα στους ερχόμενους μήνες να πιστεί και να κοιτάξει να τα αποφύγει. Έχω μια-δυο ερωτήσει, διότι μπορεί ε, σε σε επίπεδο δεν υπάρξουν αλλαγέ στο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη το γεγονό ότι δύο πράγματα μου έρχονται κατά νου. Το Βιετνάμ, ιδίω τώρα με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, είναι έτοιμο να λάβει κάποια παραγωγή από την Καμπότζη και επίσης έχει ληφθεί υπόψη ότι η Καμπότζη μπορεί να ε, συσφίξει τους δεσμούς με την Κίνα βάσει τις θέσεις που έχουμε ως τώρα εμείς και επίσης τα δικαιώματα στη γη έπαιξαν κάποιο ρόλο διότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχαν σοβαρότατες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στο Ευρωκοινοβούλιο για την λεγόμενη ζάχαρη που παράχθη, ε, παρέχθη εις βάρος του ντόπιου πληθυσμού οι οποίοι ήταν ε, όλοι απασχολούμενοι στην παραγωγή ζάχαρης. Ευχαριστούμε πάντως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, τόσο διεξοδική παρουσίαση. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μας ενημερώσει με θετικές εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μια άλλη χώρα της περιοχής, την Μιανμάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όντως είναι ατυχές που γίνεται η συζήτηση αυτή διότι ακούσαμε τον Επίτροπο Χόγκαν και ακούσαμε και το σκεπτικό του είπατε προσώπου του κ. Μπορέλ. Συμφωνώ και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει δράση και δυστυχώ χρειάστηκε να αναλυθεί. Εδώ η ουσία είναι ότι ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και θα πρέπει να είναι μη διαπραγματεύσιμο ε, στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα θα πρέπει να δούμε πραγματικέ αλλαγέ ε, στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Καμπότζη η ελευθερία του συνασπίζεστε, της έκφρασης, τα δικαιώματα στη γη, κατοχή γη και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα βασικά μάλλον δικαιώματα, είναι ε, στοιχεία που γραφίζονται διαρκώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι Καμποτζένε αρχέ είχαν κάθε ευκαιρία για να αλλάξουν τι θέσει του. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίζει την ε, έντονη προσπάθεια να είναι σε συνομιλία με τι αρχέ τη Καμπότζη και να παρακολουθεί ε, στενά το τι μέτρα μπορούν να αναλυφθούν. Ελπίζουμε να έρθουν θετικότερε εξελίξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερο εμπορικό προορισμό ε, για την Καμπότζη και η διακοπή ε, στην αποστολή προϊόντων όπω τα υποδήματα ή τα κλειστοδουλικά είναι πρόβλημα για τα ενδύματα είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι οι προγραφικές μας γραμμές, ποια όρια θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιοι πλήττονται περισσότερο εδώ. Οι καταστάσεις αυτού του είδους πραγματικά ε, είναι λεπτές η πρόσβαση στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για κάποιον ε, στην ε, Καμπότζη. Μπορεί να μείνει άνεργος λόγω της πρόσβασης αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να προκαλέσει αλλαγές στη στάση της ε, Καμποτζιανής πλευράς. Αναγνωρίζουμε όμως ότι αυτή η λύση εσχάτου καταφυγίου ήταν καλή και ήταν μια προειδοποίηση για άλλε χώρε ε, που εξηγεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν χρειαστεί, θα λάβει, αναλάβει δράση για την πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τον Πολύ σύντομα, η ομάδα μα υποστηρίζει τη γραμμή τη Επιτροπή, τη γραμμή του εισηγητή και δεν διαφωνεί με τα εξοδότηση πράξη. Δύο πολύ σημαντικοί είναι οι λόγοι. Βεβαίω η κατάσταση στην Καμπότζη και Εάν δεν το κάνουμε, θα πλήξει το σύστημα των ε, σχετικών συμφωνιών που έχουμε, Everything But Arms, και τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Και εδώ ε, το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει, έχουμε εδώ εκπροσώπηση από την Καμπότζη, τον πρέσβη. κοιτάξτε, θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη για τη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κάνουμε αυτό όχι με ενθουσιασμό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που εργάζεται στον τομέα παραγωγής ενδυμάτων, υποδημάτων. Είναι σημαντικό. Θέλουμε οι ζωές τους στην Καμπότζη να βελτιωθούν, όχι να χειροτερέψουν. Πηγαίνετε το μήνυμα πίσω στη χώρα σας. Αλλάξτε την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη, ότι εν τέλει να μην επιβληθεί αυτή η πράξη. Επόμενος ομιλητής η κυρία Σβένιαν δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα και είναι επικεφαλής αυτού του, αυτού θέματος εκ μέρους της ΡΙΝΙΟΥ. Ευχαριστώ την α, Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για την παρέμβασή τους. Ε, διαβάζω την ε, ανάλυση της ε, συναδέλφου. Ευχαριστούμε την Κομισιόν και συμφωνούμε με τη μερική αποχώρηση των προτιμησιακών δασμών. Η κατεξακολούθηση παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το δικαίωμα και την ε, πολιτική συμμετοχή, την ελευθερία έκφραση, το δικαίωμα του συνέρχεσαι και συνεταιρίζεστε από το καθεστώ τη Καμπότζη δεν μα άφησε άλλη δυνατότητα. Το καθεστώ ε, όλα πλην των όπλων και το GSPS δεν είναι δώρο, είναι μια σύμβαση με μια αναπτυσσόμενη χώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτιμησιακέ ε, ε, προτιμησιακούς δασμούς υπό τον όρο ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα και τις σχετικές συμβάσεις. Η Καμπότση όμως δεν ε, σεβάστηκε τα δικά της, το δικό της κομμάτι. Είναι η τελευταία μας καταφυγή αυτή αλλά είμαστε στην περίπτωση της Καμπότση υποχρεωμένοι να φτάσουμε στα άκρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει ότι δεν θα διστάσει να κάνει το παν για να σεβαστούν οι υπόλοιποι τις αξίες της σε περίπτωση που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσωπικά θα ήθελα να συμφωνήσω με τη δήλωση της συναδέλφου και των προλαλισσάντων συναδέλφων γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει στεναρότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η θέση θα πρέπει να είναι ένας μοχλός για να βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα. Ευχαριστώ. Ο κ. Λατσίνη. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Λαντσίνη. Να τονίσω και κάτι άλλο. Για το ρίσι ε, πήραμε μια απάντηση, μερική έστω. Το θέμα επίσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θέλω να κάνω παραλληλισμούς, αλλά νομίζω ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και για το Βιετνάμ. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι συζητήσιμο. Δεν νομίζω ότι είναι τα καλύτερα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχουμε δύο ταχύτητες, δύο μέτρα και δύο ε, σταθμά στις εμπορικές μας σχέσεις. Ε, ενώ στην πραγματικότητα είναι αντίστοιχες οι σχέσεις, αντίστοιχες οι καταστάσεις με, του Βιετνάμ με την Καμπότζη. Και τώρα ο πρέσβης έχει το λόγο για τρία λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παραστώ εδώ. Ε, ακούσαμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ τους αξιότιμους ευρωβουλευτές της Επιτροπής για την, ε, που εξέφρασαν. Ξεκινάει τώρα η επίσημη διαδικασία ε, για το EBA για την Καμπότζη. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ καλή συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καμπότζη για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα και αστικά δικαιώματα επίσης. Κάναμε ως κυβέρνηση πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει και το έχει αναγνωρίσει όλα αυτά που κάναμε μέχρι στιγμή. Στις 12 Φεβρουαρίου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εισαγάγει τη μερική αναστολή του EBA για την Καμπότζη. Η κυβέρνηση της Καμπότζης λυπάται για την απόφαση αυτή. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λάθος αντίληψη, παρανόηση για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στη χώρα μας. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ε, απτή πρόοδο που έχει γίνει σε πάρα πολλούς τομείς. Αλλά δεν αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, είναι θέματα που αποφασίζονται ανεξάρτητα ε, από τη χώρα αυτή. Για τις προτιμησιακές πρακτικές Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίω αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία το Φεβρουάριο πέρυσι. Έκτοτε έχουμε έρθει σε επαφή σε τεχνικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φτάσαμε και μέχρι το πολιτικό επίπεδο. Μιλήσαμε για τις ανησυχίες της Κομισιόν και σε όλα τα πράγματα που μας ρώτησε η Κομισιόν, απαντήσαμε ακόμα και στις τελευταίες ερωτήσεις που εκφράστηκαν στις 12 Δεκεμβρίου του 2019. Τι κάναμε στο μεταξύ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να απαντήσουμε στις ανησυχίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τις ε, νομικές διαδικασίες, δηλαδή τις διαδικασίες ενώπιων, ενώπιον ε, ε, δικαστηρίων που πρέπει να γίνουν με, τη δική τους, με το δικό τους ρυθμό. Δεν θέλουμε να προβούμε σε καμία δράση η οποία θα υποσκάψει βεβαίω την κυριαρχία μα και την ελευθερία μα. Κάτι που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι είμαστε ελεύθεροι και κυρίαρχοι. Αναγνωρίζει ότι έχουμε κάνει σοβαρή πρόοδο στο να αντιμετωπίσουμε επίσης τις ελλείψεις μας. Όλα όσα έχουν γίνει μέχρι, στιγμή, μέχρι στιγμής έχουν γίνει σοβαρά και καλή την πίστη. Με βάση τη διαδικασία που μας έχει δεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης είχαμε και το πολιτικό θάρρος να κάνουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Η απόφαση που πήρε στις 12 Φεβρουαρίου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λυπεί και έχει σοβαρότατες συνέπειες. Ανεξάρτητα από την απόφαση, εμείς ως κυβέρνηση είμαστε διατεθειμένοι για να συνεχίσουμε το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα πνεύμα αμοιβαίου συμβασμού και λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία μας συμφέροντα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι είμαστε ανοιχτές και πολυμερείς δημοκρατίες. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Ελπίζω να έρθετε να επισκεφτείτε την Καμπότζη κάποια στιγμή, να ξοδέψετε λίγο χρόνο στη χώρα μας αυτή, να δείτε και να ζήσετε και να βιώσετε τις πραγματικότητες της χώρας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πίτερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους αδελφούς για την υποστήριξη. Μια-δυο ερωτήσεις ε, τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα για το Βιετνάμ βεβαίως το σώμα σας έχει εγκρίνει προσφάτως την ε, συμφωνία RTA και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων με το Βιετνάμ. Όμως μετά από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις και συζητήσεις εσωτερικός και σε συνεργασία με το Βιετνάμ ε, την ίδια μέρα συμπτωματικά ενέκρινε και το κολέγιο των επιτρόπων την ε, άρση την αναστολή των τη προτιμησιακή μεταχείρισης για την Καμπότζη. Βεβαίω ξέρετε ότι είναι διαφορετικά εργαλεία αυτά. Δηλαδή, κοιτάζουμε να γίνονται σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα. Ε, η το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων δίνει μονομερώς βάση προϋποθέσεων κάποια ευνοϊκή πρόσβαση, ενώ η συμφωνία FTA είναι διαφορετικού είδους και εντοπίζεται μεν στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά σε εταιρικέ σχέσεις με διάσταση, με συνιστώσεις για το περιβάλλον, ε, πράγματα που τα βλέπουμε στι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Και τα δύο είναι εργαλεία για να βελτιωθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών και να μπορούμε να δούμε και την κατάσταση στην κάθε χώρα. Βλέπουμε και υπήρξαμε μάρτυρε αυτού ότι υπάρχουν σοβαρέ προσπάθειε από την πλευρά του Βιετνάμ και από την πλευρά τη Καμπότζη για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση σε ό,τι αφορά το να λάβουμε υπόψη το πώς θα επηρεάσει η Συμφωνία Ελευθερών συνελεγών με το Βιετνάμ και πώς θα υπάρξει αναστολή των γενικευμένων υποτιμήσεων για εταιρείε που ούτως ή άλλως έχουν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον ενό έτους για τη λειτουργία του. Ήρθαμε σε επαφή με εταιρείε που ήρθαν, μας παραπονέθηκαν, μα είπαν τα προβλήματά τους. Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν σαφήνεια, να είναι κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Πρέπει να ξέρουμε πώ θα δημορφωθεί η κατάσταση. Όμω εν τέλει είναι. Ε, θέμα προτίμησης και πολιτικής, το αν θέλουμε να στείλουμε ε, παραγγελίες σε χώρα με τις οποίες έχουμε μονομερώσεις προτιμήσεις ή συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, τώρα με την Κίνα. Το πόσο πιο κοντά θα πάμε είναι ένα θέμα. Πάντως, οι εμπειρογνώμονες της Καμπότζης έρχονται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε φοβεροί εταίροι για την Καμπότζη και ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ως προς την αρπαγή γεών και τα δικαιώματα κατοχής γης. Είδαμε, ε, και το λέει και η πράξη μας, ότι έχει γίνει σοβαρή πρόοδος στην επίλυση διαφορών ε, κατοχής γης. Οι ΕΛΣΙΣ λέγονται με τις λεγόμενες υποχρεωτικέ παραχωρήσεις. Για την ε, ζάχαρη, από τότε που αναλύθη η δράση μας, υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, τυπλοποίησης ε, οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν με μια αμερόληπτη και ουδέτερη εφαρμογή προς το όφελος των ηθαγενών πληθυσμών. Πολλά έχουν εξαλειφθεί και είναι φυσικό ότι αυτά θα οδεύσουν προς λύση όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πιέζουμε την κυβέρνηση της Καμπότζης για να το κάνει γρήγορα. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας, Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μάριος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε ουσιαστικά σε όλα τα ερωτήματα, οπότε δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ω, έκπληξη, λέει ο Πρόεδρος. Συνήθως δεν συμβαίνει, συμβαίνει το αντίστροφο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε, ολοκληρώνεται το θέμα 14 και κάνω ένα, μια σύντομη διακοπή ενό λεπτού. Το επόμενο θέμα ε, θα συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Και άρα όποιος δεν δικαιούται να παραμείνει στη συζήτηση αυτή και κλεισμένο των θυρών θα πρέπει να φύγει ησύχως.